Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε την ε, συνεδρίασή μας και βρισκόμαστε στο σημείο 21 της ημερήσιας διάταξης. Νέα μεθοδολογία για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων ε, εκ μέρους τρίτων χωρών. Είναι Σημαντική αυτή η νομοθεσία. διότι σε όλο τον κόσμο βλέπουμε όλο και περισσότερα προϊόντα dumping και παράνομα επιδοτημένα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τη βιομηχανία μας. Γι' αυτό εδώ και αρκετό καιρό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει σχετική πρόταση. Ιδιαίτερα μία μεγάλη χώρα προκαλεί προβλήματα που επί 15 χρόνια 15 ε, ε, ε, χρόνια διήρκησε η διάρκεια προσχώρησης της στον ΠΟΕ. Τώρα λοιπόν έχουμε τη σχετική νομοθεσία και και είναι ασυνήθιστο αυτό, ε, έχει γίνει αντικείμενο επίθεσης αυτή η νομοθεσία, παρότι δεν είναι καν έτοιμη ακόμα. Έχουμε λοιπόν μία υπόθεση στη Γενέβη, στον ΠΟΕ, ε, από πλευράς της Κίνας, ε, που έχει προσφύγει κατά της παλαιάς, αλλά και αυτής της νέας νομοθεσίας που δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ και άλλα μέλη του ΠΟΕ φαίνεται να στηρίζουν αυτό το αίτημα της Κίνας, ε, η Ινδονησία, οι χώρες του κόλπου, η Ρωσία και άλλοι. Πολιτικά λοιπόν είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Και αυτό αναγνωρίστηκε και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο λοιπόν χθες υιοθέτησε εντολή διαπραγματευτική με το Κοινοβούλιο. Ενήργησε λοιπόν πιο γρήγορα το Συμβούλιο αυτή τη φορά και γι' αυτό το λόγο έχω καλέσει το Συμβούλιο να παρουσιάσει και τη δική του θέση εδώ σήμερα, αλλά φυσικά μετά από τη δική μας συζήτηση. Η δική μας συζήτηση θα ξεκινήσει με την εισαγωγή του εισηγητή μας. Του δίνω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι τα όσα είπατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Ε, όλα αυτά οδηγούν σε πολύ σημαντικούς προβληματισμούς και σκέψεις. Ε, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Στις 9 Νοεμβρίου του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία πρόταση ε, η οποία πραγματοποιεί τροποποίησεις ε, στη στάνταρ μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαδικασίες αντι-dumping και κατά των επιδοτήσεων. Στην πρόταση αυτή ε, αυτή η πρόταση είναι συμπληρωματική όσον αφορά τα εργαλεία ε, υπεράσπισης του εμπορίου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση στον τριμερή διάλογο μεταξύ Συμβουλίου, ε, Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν υποτίθεται ότι είναι ουδέτερη όσον αφορά τις χώρες, country neutral. με κάποια διαφοροποίηση μεταξύ χωρών που είναι οικονομίες αγοράς και χώρες που δεν είναι. εφαρμόζεται ισότιμα σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές τρευλώσεις της αγοράς όπως ε, καθορισμός των τιμών. Η μόνη διαφοροποίηση που έχει απομείνει αφορά τις χώρες μέλη του ΠΟΕ και τις χώρες μη μέλη του ΠΟΕ για τις οποίες χρησιμοποιείται το ε, σύστημα χώρας ανάλογης με οικονομία αγοράς. Η πρόταση αυτή είχε την πρόσφατη προθεσμία του πρωτοκόλλου 16 της προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ. Στο πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει στα μέλη του οργανισμού να χειρίζονται την Κίνα ως χώρα που δεν έχει οικονομία αγοράς. Έτσι λοιπόν οι δασμοί αντι-dumping υπολογίζονται εφαρμόζοντας μια εναλλακτική μεθοδολογία αντί για τη στάνταρ μεθοδολογία. Ως αποτέλεσμα της προθεσμίας ε, της παραγράφου 15αε ε του πρωτοκόλου προσχώρησης των ε, ΠΟΕ της 12 Δεκεμβρίου του 2016 η Κίνα ζήτησε για τις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ορισμένες διατάξεις του κοινοτικού κανονισμού που σχετίζονται με τον καθορισμό της κανονικής αξίας για τις χώρες που δεν είναι οικονομίας αγοράς, τις διαδικασίες αντι-dumping, όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα. Και όπως υπενθυμίσετε και εσείς κύριε Πρόεδρε, η Τσίνα επισημοποίησε το Μάρτιο του 2017 μία προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζετε. Από τότε που δημοσιεύτηκε η πρόταση της Κομισιόν, οι αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι αντιδράσει του Κοινοβουλίου ε, υπήρξαν μεγάλες ε, φόβος, ε, αβεβαιότητα ε, μία ε, στάση που εμείς ε, θεωρούμε κατανοητή. Οι αντιδράσεις αυτές, ωστόσο, μας κάνουν να συνειδητοποιούμε ότι είναι αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους του ΠΟΕ. Ε, ταυτόχρονα όλα αυτά γίνονται σε εποχές ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές, αρκετά περίπλοκες. Ε, σε τέτοιες εποχές η βιομηχανία μας, όπως ξέρουμε, ε, πλήττεται από μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση και από τις προκλήσεις που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση. Όπως σας είχα ήδη ανακοινώσει, θεωρώ ότι είναι ύψης της προτεραιότητας να κάνουμε μια σειρά αναλύσεων. Μαζί σας, Πρόεδρε, είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους εκπροσώπους του δικού μας ε, Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Συστήματος των ε, ενώσεων ε, που μας παρουσίασαν τη δική τους εικόνα βάσει της δικής τους εμπειρίας, των ικανοτήτων τους, των δυνατοτήτων τους για την υπεράσπιση ενός συστήματος το οποίο πολύ συχνά τους τιμωρεί. Θεώρησα όμως εγώ ότι ήταν απαραίτητο να συναντήσουμε και τους Αμερικανούς μας εταίρους γιατί ήθελα να γίνει μια συγκριτική ανάλυση, να δούμε σε σχέση με το δικό του σύστημα τι συμβαίνει. Επειδή το δικό του σύστημα ούτω ή άλλω είναι ένα μοντέλο αναφορά ε, και διασφάλιση τη προστασία τη Αμερικανική βιομηχανία. Το λέω λοιπόν ενημερωτικά προς τους συναδέλφους. Επισκέφθηκα ε, ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συνάντησα εκπροσώπους της βιομηχανίας απευθείας ε, των διαφορών χωρών, των χωρών που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδα ποια είναι η εικόνα της βιομηχανίας μας σε όλους τους τομείς, ειδικότερα όσοι πλήττονται από το ντάμπινγκ, ο χάλιβας, τα κεραμικά, τα ποδήλατα, τα φωτοβολταϊκά, ε, το χαρτί και όλα τα παράγωγα προϊόντα. Κατά τη σύνταξη του σχεδίου που σας παρουσιάζω σήμερα, ακολούθησα μία μέθοδο την οποία θεώρησα ιδανική για την επίτευξη τριών σκοπών. Πρώτον, προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υπεράσπιση της, η οποία ενώπεν όλων των προγραμμάτων και των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί και από την Ευρώπη, από τον κύριο Γιούνκερ στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020, θα έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στις διεθνείς αγορές και δεδομένη τώρα της ε, υπερβολικά, ε, του υπερβολικού προστατευτισμού του Τράμπα και των συνεπειών του Brexit ε, ειδικότερα τώρα στο πλαίσιο της αντιπαρατησής με την Αγγλία. Δεύτερος σκοπός να ενσωματωθεί η, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να αλλάξει η φύση της. Γιατί, διότι εμεί κινούμαστε σε ένα χώρο πολύ ευαίσθητο νομικά και νομοθετικά. Πρέπει να προστατεύουμε και να παρέχουμε εγγυήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά το σύστημα των βιομηχανιών μας, αλλά πρέπει να προστατευτούμε ε, και σε σχέση με αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, την ανησυχητική Κίνα ε, και τις άλλες χώρες που προκαλούν ανησυχίε, ε, τις άλλες χώρες που θα μπορούσαν να προσφύγουν ε, ε, εν τέλει σε μια τέτοια πρόταση. Αυτή η πρόταση λοιπόν θα πρέπει να μας καταστήσει συμμορφούμενους με τους διεθνείς υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΕ. Δύο βάσεις λοιπόν ε, ε, ισχυρές ε, όπου πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα και συνείδηση. Θεωρώ ότι μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η προστασία του δικού μας ρόλου, του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν για Πολλέ φορέ, ε, θέλοντα να αναθεωρήσουμε αυτή την πρόταση τη Κομισιόν αναφέρομαι στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κίνα ειδικότερα εκείνη του περασμένου Μαΐου. Δεν χρειάζεται να το υπενθυμίσω, το έχουμε υπενθυμίσει πολλές φορές. Είμαστε συνομοθέτες. Είμαστε δηλαδή ε, ισότιμος εταίρος, ε, βασικός εταίρος με πολύ συγκεκριμένο ρόλο, τον οποίο δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε σε άλλους. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, η μέθοδος εργασίας ε, επικεντρώθηκε σε ορισμένες βασικές πτυχές ε, που θεωρώ ότι είναι ύψης της σημασίας. ώστε να συμμετέχουμε επικοδομητικά στις εργασίες της Κομισιόν. Ε, χρησιμοποιώ λοιπόν συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να ορίσουμε τις τρευλώσεις. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το βάρος της απόδειξης, ο ρόλος του Κοινοβουλίου, όλες οι πτυχές δηλαδή που αναγκαστικά για μένα και για τους συναδέλφους με τους οποίους συζήτησα, τους εισηγητές δηλαδή των διαφόρων κομμάτων, ε, των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου μας, ε, επιτελεί και όλο αυτό και κάποια, καλύπτει και κάποια ανάγκη και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό για τους συναδέλφους. Να υπογραμμίσουμε λοιπόν ε, την ε, απουσία διάκρισης ε, μεταξύ της Κίνας πριν και της Κίνας τώρα. εγώ το πράττω αυτό για να καταλάβουμε ότι για τις σημαντικές στρεβλώσεις απαιτείται να, εφαρμοστεί το άρθρο αυτό που αναφέρεται από την Επιτροπή αυτή και όχι απλά να αναφέρουμε ξεχωριστά τα κριτήρια στρέβλωσης. Να ενταχθεί δηλαδή αυτό το άρθρο στην νομοθεσία ώστε να μην κάνουμε το σφάλμα, να αφήσουμε περαιτέρω ευκαιρίες ανοιχτές ε, από τεχνική άποψη ή από νομοθετική άποψη τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν οι χώρες που αναφέρατε εσείς ε, συμπεριλαμβανομένες της Κίνας γιατί ξαφνικά γινόμαστε, κάνουμε μια διάκριση της Κίνας ε, εκτός του ΠΟΕ και εντός του ΠΟΕ. Ε, θέλουμε δηλαδή να δώσουμε έναν ορισμό στις τρευλώσεις που αφορούν τους διάφορους τομείς ε, όπου χρειάζεται προστασία η βιομηχανία μας. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν εισάγει αυτόν τον όρο σημαντικές τρευλώσεις για να αναφερθεί σε τι. Στις συνθήκες υπό τις οποίες οι τιμές και τα εσωτερικά κόστη δεν αποτελούν λογική βάση για να αξιολογηθεί η σωστή τιμή ενός αγαθού και η αξία του. Για να εφαρμόσουμε τη νέα μεθοδολογία πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει ε, σημαντικές στρεβλώσεις διότι από αυτές θα εξαρτηθεί η εφαρμογή της νέας μεθόδου. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε και να ενσωματώσουμε το 2.6β ε, σε περίπτωση που, υπάρχουν, που πληρούνται οι συνθήκες που θεωρούνται απαραίτητες ε, για να διαπιστωθεί η παρουσία αυτών των στρεβλώσεων. Πρώτη πτυχή, απουσία ε, διαφανούς ε, δικαίου για τις επιχειρήσεις, απουσία ε, καθεστώτος λειτουργικού, ε, μισθολογικές συνθήκες που δεν απορρέουν από συμφωνίε ε, με συνδικαλιστικές οργανώσει και οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που μπορεί να τεκμηριώσει σημαντικές τρευλώσει. Τώρα για την έκθεση, το report, ε, το θεώρησα το κεντρικό σημείο, ε, τον πυρήνα του κανονισμού αυτού. Γιατί, διότι μέσω της έκθεσης αναπτύσσουμε στη συνέχεια και την έννοια του βάρους της απόδειξης και αναπτύσσουμε επίσης και την έννοια της ε, δυνατότητας υπεράσπισης και ε, διασφάλισης ε, της βιομηχανίας μας. Θεώρησα λοιπόν ότι η έκθεση θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ειδικότερα σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει μια αρχή που να έχει τη διακριτική ευχέρεια. Η έκθεση λοιπόν δεν μπορεί, πρέπει να δημοσιεύτει ωστόσο με λεπτομερή τεκμηρίωση που να περιγράφει τη συγκεκριμένη κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χώρα και στον κάθε τομέα στον οποίο αναφερόμαστε. Όχι λοιπόν με, γενικό, με γενικόλογη διατύπωση, να αναφέρεται στους συγκεκριμένους τομείς που αποτελούν το αντικείμενο της αντιπαράθεσης μεταξύ της δικής μας βιομηχανίας και της βιομηχανίας των άλλων εξαγωγικών χωρών η δική μας ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ε, έκθεσης ώστε να υπάρχει μια παρακολούθηση, μια επαλήθευση, ένας έλεγχος, η δυνατότητα για τη βιομηχανία μας να εντοπίσει και τα διάφορα αδύναμα σημεία. Όπως είπα πριν υπάρχει το βάρος της απόδειξης, διότι ξέρετε αρχικά Όλοι θεωρήσαμε ότι έτσι όπως έχει συνταχθεί η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, ουσιαστικά αντιστρέφει την κατάσταση, δηλαδή από τη σημερινή κατάσταση, από το σημερινό κανονισμό βάση, όπου η δική μας βιομηχανία εξαιρείται απόλυτα από οποιοδήποτε, οποιαδήποτε υποχρέωση να παρέχει ε, αποδεικτικά στοιχεία, περνάγαμε σε μια κατάσταση αντιθέτως όπου υπήρχε αυτό το βάρος της απόδειξης για μας. Οπότε εγώ θεώρησα ότι στο άρθρο 2, παραγραφός 6β, ε, ε, εδάφιο D, εάν τα συμπεράσματα της έκθεσης καταδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων, η ίδια η έκθεση αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο βέβαιο, το οποίο τεκμηριώνει το, ε, ότι είναι απαραίτητο να γίνει ο υπολογισμός βάσει της νέα μεθοδολογία. Και σε κάθε περίπτωση αυτό το περαιτέρω βάρος απόδειξης ε, βαρύνει την βιομηχανία της Ένωσης. Όπως είπα, δεν πρέπει να έχουμε κανένα επιπλέον βάρος απόδειξης για τη δική μας βιομηχανία. Δηλαδή η Κομισιόν αναλαμβάνει το βάρος του να προσδιορίσει εάν σε κάποιο τομέα και στην αξιολόγηση των συστημάτων των διαφόρων χωρών με τα κριτήρια στρέβλωσης τα οποία εμείς έχουμε διευρύνει και ενσωματώσει με μία έννοια λοιπόν που θωρακίζει και επιτρέπει στην Κομισιόν να παρέχει πραγματική προστασία στο δικό μας ε, σύστημα ε, βιομηχανιών. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εμείς ε, με κάτι τέτοιο μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτό που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα πραγματοποιεί καμία διάκριση μεταξύ χώρας με οικονομία αγοράς και χώρας χωρίς οικονομία αγοράς αλλά ταυτόχρονα με αυτή την έννοια της σημαντική τρέβλωσης και την έκθεση η οποία αποτελεί στοιχείο το οποίο εξαιρεί τη δική μας βιομηχανία από το βάρος απόδειξης πληρείται στο τέλος η συνθήκη αυτή, ε, έτσι το πιστεύω εγώ και σας ζητώ συνάδελφοι να με βοηθήσετε σε αυτόν τον προβληματισμό διότι θεωρώ ότι και στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο που ξέρουμε θα είναι πολύ ευαίσθητε και λόγω των θέσεών του θα έχουμε ε, πολλά να συζητήσουμε. Ε, τώρα, για το ρόλο του Κοινοβουλίου, τέλο, ε, αυτό ο ρόλο ε, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την άποψή μου στην παρούσα φάση για αυτού του είδου τι ε, καταστάσει. Για το άρθρο 2, λοιπόν, παράγραφο 6β, ε, και εδάφιο C, ε, συγγνώμη, εκεί θέλησα να συμπληρώσουμε το κείμενο με κάποιες τροπολογίες ε, όπου το Κοινοβούλιο θα ε, αποτελεί τον εγγυητή των συμφερόντων της βιομηχανίας και των Ευρωπαίων πολιτών και γι' αυτό έτσι έχω αλλάξει το άρθρο ως εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί την εκπόνηση της έκθεσης μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπτωση αλλαγής των συνθήκων σε μια συγκεκριμένη χώρα ή τομέα, η Κομισιόν επικαιροποιεί την έκθεση. Σε κάθε περίπτωση η Κομισιόν προβαίνει σε αναθεώρηση της έκθεσης κάθε δύο χρόνια. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με την Κομισιόν όσον αφορά το ζήτημα της ανάγκης να προβλεφθεί μία μεταβατική περίοδος μεταξύ της κατάργησης της εφαρμογής του σημερινού ε, κειμένου βάση προς όφελος του κειμένου που εμείς συζητάμε σήμερα και το οποίο πρόκειται να ψηφίσουμε. Θεωρώ πράγματι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ότι μέχρι σότου εφόσον οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει στους εξαγωγείς που αναφερόμαστε ε, εφόσον διαπιστωθεί ότι ε, το επίπεδο των δασμών δεν είναι επαρκές και ε, εφόσον πρέπει να γίνει επανυπολογισμός βάσει της παλιάς μεθοδολογίας η πρόταση αυτή θεωρώ εγώ ότι δεν θα πρέπει να, να τροποποιηθεί διότι προστατεύει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα της δικής μας βιομηχανίας να μπορέσει να επιβιώσει για κάποιους μήνες, κάποια χρόνια υπό καθεστώς μεγαλύτερης ακόμη προστασίας. Ε, ε, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστώ ίσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συμβολή τους και φυσικά απομένουν πολλά να γίνουν από εμάς και αναμένω τις σκέψεις και τα σχολιά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την εντατική δουλειά που κάνατε πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε περιορισμένο χρόνο να συζητήσουμε γιατί θέλουμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τη δήλωση του Συμβουλίου. Συνεπώς, προτείνω 2,5 λεπτό καθένας. Θα αρχίσω με τους σκιώδεις εισηγητές, εννοείται. Πρώτα από τους σοσιαλιστές, Εμμανουέλ. Ευχαριστώ. Έχει δίκιο ο συντάκτης που αναφέρει και επαναλαμβάνει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί πρέπει να είμαστε πράγματι πάρα πολύ προσεκτικοί εδώ, να είμαστε αποφασιστικοί και να βάλουμε ψηλά τον πύχη. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και οι εξελίξεις στο Συμβούλιο είναι μάλλον απογοητευτικά πράγματα σε σχέση με τις φιλοδοξίες μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, ε, σε αντίθεση με τους εταίρους μας, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Βραζιλία κτλ, δυσκολεύονται να βρούνε ένα σύστημα για να προστατευτούν και να προστατεύσουν τις βιομηχανίες τους. Και εμείς έχουμε μια τέτοια δυσκολία βέβαια. Λοιπόν, με την έκθεση Τσίκου και με τα όσα μπορούμε να κάνουμε όλοι, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση και να βάλουμε όλα τα στοιχεία αποφασιστικότητας που χρειάζονται προκειμένου να προστατεύσουμε την Ευρώπη καλύτερα, γιατί σήμερα δεν προστατεύεται αποφασιστικά. Σύμφωνοι για τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην οικονομία της αγοράς και τη μη οικονομία της αγοράς, αλλά αν πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση, τότε να ενισχύσουμε τη μεθοδολογία anti-dumping που χρησιμοποιούμε. Πρώτον, λοιπόν, μια που μας ζητήσατε να είμαστε γρήγοροι, σύντομοι. Πρώτον, λοιπόν, το κείμενο δεν πρέπει να αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης. Δεν είναι οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν κάτι. Όχι, οι Κινέζοι πρέπει να το αποδείξουν. Δεύτερον, το είπε και ο εισηγητής, η έκθεση με το νέο σύστημα. Κάθε νέα μεθοδολογία δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αν δεν υπάρχει αυτή η έκθεση. Αλλά η έκθεση θα πρέπει να είναι πολύ απαιτητική και όσον αφορά την έκθεση, και την ποιότητά της και όσον αφορά τη δομή της γιατί έχουμε μια μεθοδολογία που δεν είναι στάνταρτ. Και τρίτον, πιστεύω ότι πρέπει να επεκτείνουμε τον κατάλογο των ε, παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή τη σημαντική στρέβλωση, σε σημαντικές στρεβλώσεις. Δεν είναι προσυζήτηση σήμερα αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Να προσθέσουμε κριτήρια. Κριτήρια που μπορούμε να βρούμε στο Αμερικανικό δίκαιο, αλλά επιπλέον να βάλουμε κοινωνικά κριτήρια, περιβαλλοντικά κριτήρια. Και τρίτον, Νομίζω ότι πρέπει να προβλέψουμε και μηχανισμούς κύρωσης αν δεν υπάρξει συνεργασία του εξαγωγέα όταν λαμβάνει η χώρα η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες αυτές οι διατάξεις εμπνέονται από τη σχετική νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να τυχαίνουν τις ίδιες μεταχείρισεις όπως οι μεγάλες βιομηχανίες, γιατί είναι οι πιο εύθραυστες σε μια κατάσταση dumping. Μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά πρέπει να βάλουμε τον πύχη πιο ψηλά από ό,τι βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, βέβαια, γιατί ξέρουμε ότι το Συμβούλιο δεν είναι στο ύψο που πρέπει. Ευχαριστούμε. Λούνε από το ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και τον ε, εισηγητή για το κείμενό του που πιστεύουμε ότι είναι μια επικοδομητική προσέγγιση που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και σίγουρα είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να δουλέψουμε παρετέρω. Υπάρχει ευρεία συνένεση ότι πρέπει να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό που βασίζεται σε κανόνες, μια ανοιχτή επίσης αγορά, μια ελεύθερη αγορά. Για την ομάδα μας, για το ECR, είναι ζωτική σημασία να έχουμε ένα σύστημα που θα διασφαλίζει την ίδια αποτελεσματικότητα βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, όπως υπόθηκε. Συγχρόνως είναι σημαντικό για μας να λάβουμε υπόψη μας το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή και η ποιότητα, αλλά η ποιότητα συνδέεται και με το χρονοδιάγραμμα. Οι στόχοι του εισηγητή μας βρίσκουν σύμφωνος, δηλαδή η μεθοδολογία έτσι ώστε να μην είναι τόσο δύσκολος ο υπολογισμό ε, του dumping Δεύτερον, ο μηχανισμός να είναι πιο αποτελεσματικός για την καταπολέμηση του dumping και να μην μπαίνει επιπλέον βάρος στις επιχειρήσεις μας, κυρίως, όπως είπε και ο σκέτος ηγητής των σοσιαλιστών, στις μικρομεσαίες. Τώρα, για τις σημαντικές τρευλώσεις. Εδώ θέλω να, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, ο οποίος πράγματι διευκρινίζει περισσότερο το τι σημαίνουν οι σημαντικές ε, στρεβλώσεις και πώς ε, εξηγεί αυτόματα θα χρησιμοποιούμε τις τιμές της αγοράς. Για τις εκθέσεις, ναι, συμφωνούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι πρέπει να εκδίδει έκθεση κάθε φορά που εντοπίζονται σημαντικές τρευλώσεις. Αναρωτιόμαστε βέβαια για το ρόλο του Κοινοβουλίου, στην πράξη δηλαδή και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί η έκθεση λέει ότι θα ελέγχει τη διαδικασία σύνταξης της έκθεσης. Στην πράξη πώς θα γίνει όμως αυτό, αναρωτιέμαι. Είναι μια ανάλυση που γίνεται βάση στοιχείων, οπότε πώς ε, εμπλέκεται εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επιπλέον έχουμε και μια πρόταση. Ο εισηγητής συζητάει μια προέκθεση. Είναι καλή πρόταση εμείς θα λέγαμε να είναι υποχρεωτικές οι εκθέσεις αυτές για τις χώρες εκείνες για τις οποίες έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αξιολόγηση στο παρελθόν. Κίνα, αλλά και Αρμενία για παράδειγμα. Βάρος της απόδειξης τώρα. Για το βάρος της απόδειξης συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το μηχανισμό αυτό. Το βάρος της απόδειξης παραμένει με την πλευρά των εκείνων που προσφεύγουν, έτσι, οπότε προσοχή. Τώρα για το αμερικανικό σύστημα το έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε περισσότερο από τον εισηγητή για το πώς το βλέπει αυτό το αμερικανικό σύστημα στη δικιά μας περίπτωση. Ευχαριστούμε. Λάμστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πράγματι θα μιλήσω στο όνομα του κυρίου Λάμστορφ, αλλά επιτρέψτε μου να μου δώσετε λίγο χρόνο για να σας παρουσιάσω και τις δικές μου θέσεις. Καταρχάς, ο κύριος Λάμστορφ ευχαριστεί τον εισηγητή που έχει θέσει φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό, ώστε αν όλα πάνε καλά να κλείσουμε πριν το καλοκαίρι. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το βασικό αντικείμενο αυτής της πρότασης, να αντιμετωπίσουμε τις νομικές προκλήσεις που απορρέουν από τους κανόνες του ΠΟΕ και να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αναλαμβάνει εγκαίρως αποτελεσματικά βήματα και επίσης να μην δημιουργήσουμε επιπλέον ε, άχθος για την βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Λάμστορ πιστεύει ότι το πρώτο σχέδιο είναι πολύ καλό. Απομένουν όμως αρκετά να γίνουν ακόμα. Να σας ε, αναφέρω κάποια σημεία αναφέρεται στο ότι έχει συμπεριληφθεί ένα μη εξαντλητικό κατάλογο κριτηρίων. Είναι σημαντικό ο κατάλογο αυτό να παραμείνει ανοιχτό, ώστε να υπάρχει περιθώριο για την Κομισιόν να διασφαλίζει την πιο αποτελεσματική προστασία τη ευρωπαϊκή βιομηχανία, ε, χωρί να κλείσει την ε, κοινή αγορά. Ωστόσο, όσον αφορά τα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια, θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικά τι αναφέρεται. Αμφιβάλλω, για παράδειγμα, ότι ένα καθεστώς αφαιρεγκιότητα ε, μπορεί να μας ε, πει πολλά για την παγκόσμια οικονομία που αλλάζει. Επίση, οι τιμέ τη ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ω benchmarks, διότι ήδη συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό των τιμών αναφοράς. Επίσης, οι εκθέσεις ε, αναχώρα ή ανατομέα ε, ενδεχομένως να καθυστερήσουν περαιτέρω την όλη διαδικασία, διότι ο ισχύων κανονισμός είναι ε, πολύ αποδυναμωμένος και είναι σημαντικό να μην ε, αποκρίτουμε από τις ε, βιομηχανίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε μια νομικά ισχυρή πρόταση. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η διεύρυνση του ρόλου των ενδιαφερομένων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά σύμφωνα με το κείμενο οι χώρες ε, θα είναι σε θέση να ε, σχολιάσουν την ε, έκθεση αυτή. Η έκθεση όμως θα πρέπει να είναι αντικειμενική. Επιπλέον επικροτούμε το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων δεν πιστεύουμε όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένη έκθεση. Επίσης, ε, η αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια δεν ε, μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμά, διότι αποτελεί ε, μέρος της συζήτησης ανατομέα που γίνεται σε κάθε χώρα κάθε 24 μήνες. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που προβλέπονται στο θέμα αυτό αρκούν να ζητήσω το λόγο αργότερα για τις δικές μου θέσεις. Πρόεδρος, ναι, μας τελειώνει ο χρόνος. Ήδη ξεπεράσατε το χρόνο κατά ένα λεπτό. Ε, Χέλμουντ Σόλτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλους τους συναδέρφους και ιδιαίτερα τον εισηγητή ότι πρόκειται για πολύ ε, σημαντική νομοθεσία και έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να μπούμε στα επιμέρους ζητήματα του συγκεκριμένου σχεδίου έκθεσης. Ε, τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Έχουμε μια πλήρη εργαλειοθήκη, επικροτώ την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύσουμε την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το πλαίσιο και στον τομέα του περιβάλλοντος των δικαιωμάτων κλπ. Ε, δεν θέλουμε το dumping να ε, διακυβεύει την ε, παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία θα πρέπει να συνδυάσει τις διάφορες απόψεις σχετικά με τον τρόπο καλής λειτουργίας της βιομηχανίας. Ας σκεφτούμε την Κίνα. Η Κίνα έχει άλλο ορισμό της οικονομίας της αγοράς από ότι εμείς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όταν μιλάμε για μισθούς, την κοινωνική νομοθεσία θα πρέπει πρώτον να συμμορφωνόμαστε με τον ΠΟΕ, να ακολουθούμε δηλαδή τους κανόνες του ΠΟΕ για να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας. Θα πρέπει τα επιτεύγματά μας να τα προστατεύουμε από το ντάμπινγκ και για παράδειγμα κατά την διαπραγμάτευση των μισθών, όπως λέει και η έκθεση, και είναι σωστή η διατύπωση στην έκθεση αυτή, διότι το θέμα δεν είναι οι μισθοί ε, να διαμορφώνονται ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις μας με τους ε, εξωτερικούς μας εταίρους. Ένα παράδειγμα σας δίνω, η ενεργειακή πολιτική. Για παράδειγμα, έχουμε τρόπο να παρέμβουμε στην ε, διαμόρφωση των τιμών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προστατεύσουμε τους τομείς αυτούς. Πιστεύω ότι Χρειαζόμαστε μια περίοδο προβληματισμού σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητέ για να εξετάσουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του εισηγητή και να τις επικαιροποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή ο οποίος σαφώς έχει βελτιώσει σημαντικά την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την εναλλακτική μεθοδολογία, την αυτοματισμό, το βάρος της απόδειξης, όλα αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί, διότι ε, σίγουρα η Ευρώπη έχει μεν μια κοινή εμπορική πολιτική, αλλά είναι σαφές ότι λόγω απουσίας βιομηχανικής πολιτικής δεν υπάρχει κοινή εμπορική στρατηγική ή διπλωματία και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση όπως και η έκθεση για τα εργαλεία άμυνας του εμπορίου δημιουργούμε μια κοινή στρατηγική που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις ε, dumping και την Κίνα. Το είδαμε στα φωτοβολταϊκά, στη σιδηρουργία. Υπάρχει αυτή η έλλειψη ενός ισχυρού κοινού ευρωπαϊκού και αυτό καταστρέφει την εικόνα της Ευρώπης ε, και την κατάσταση πολλών πολιτών ε, και μισθωτών. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο μας υποχρεώνει να είμαστε φιλόδοξοι. Εδώ βλέπω και τη σχέση με τα εργαλεία εμπορικής άμυνας και το σχετικό εγχείρημα. Φυσικά σε περιπτώσεις σημαντικής τρέβλωσης, ό,τι σχετίζεται με το περιβάλλον μπορεί να, και μπορεί να επηρεάσει τις τιμές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Παρομοίως, ό,τι κάνουμε, όπως κάνουμε και στα εργαλεία εμπορικής άμυνας και το είδαμε στην περίπτωση της σιδηρουργίας, είναι να έχουμε τη συμμετοχή των συνδικάτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό και πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Σε περίπτωση διαβουλεύσεων με τους βιομηχάνους καθώς χρειάζεται η αλληλεπίδραση με τους βιομηχάνους, ε, πρέπει να συμμετέχουν ε, ενεργά και τα συνδικάτα. Το είδαμε στη σιδηρουργία, όπως είπα, συμμετείχαν σημαντικά στην κινητοποίηση διάσωσης ε, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τέλος, πρέπει να καταβάλουμε κάποιες προσπάθειες όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τους εξαγωγείς, ε, υπόθηκε ήδη. Χρειάζεται να ανεβάσουμε λίγο τη φιλοδοξία τόσο εδώ στη δική μας ε, Επιτροπή ενώπιον του Συμβουλίου και της Κομισιόν, διότι για άλλη μια φορά, συζητώντας για την Ευρώπη σήμερα, είναι απολύτως αναγκαίο να είμαστε αποφασιστικοί για να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας, τους ε, εργαζομένους και τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλέσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτω με τον εισηγητή μα σε δύο βασικά θέματα. Την ανάγκη να καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιε είναι αυτέ οι σημαντικέ στρεβλώσει και να καταλάβουμε και το ρόλο των εκθέσεων και τη όλη διαδικασία. Να πω όμω κάτι για κάτι που λείπει και νομίζω θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτή η μεθοδολογία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χώρε άλλε από την Κίνα. Όπως γνωρίζετε, οι σημαντικές στρεβλώσεις, ε, έχουμε σημαντικές στρεβλώσεις σε βασικές πρωτεσίλες σε όλον τον κόσμο. Και στο παρελθόν, ε, οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, καθοριστεί σωστή τιμή για τις ύλες αυτές, οι κανόνες αυτοί βρίσκονται υπό επίκριση αυτή τη στιγμή στον ΠΟΕ. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτή η μεθοδολογία να μπορεί να ισχύσει η δική μας μεθοδολογία να μπορεί να ισχύσει σε διάφορες περιπτώσεις δηλαδή. Πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στην ανάγκη για ευελιξία και καταλαβαίνω την αφετηρία της Κομισιόν που είναι οποιαδήποτε μεθοδολογία υιοθετήσουμε να μην μας οδηγήσει σε ήττα στον ΠΟΕ, κάτι που θα σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε όλη την νομοθεσία αντι-dumping της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην χάσουμε λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει οι κανόνες μας να είναι ευέλικτοι ώστε ε, κανένας φορέας του ΠΟΕ να μην καταλήξει ότι οι κανόνες μας είναι παράνομοι σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Εάν όμως δώσουμε την ε, ευελιξία αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να περιορίσουμε τις ε, επιλογές της, όχι μόνο ενισχύουμε την θέση μας στον ΠΟΕ, αλλά χάνουμε και τον έλεγχο της Κομισιόν. Το θέμα λοιπόν είναι, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τους δώσουμε αρκετή ευελιξία και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να κάνει τη σωστή δουλειά για να εντοπίσει σημαντικές τρευλώσεις στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να σκεφτούμε στρατηγικά και μακροπρόθεσμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε περιθώριο υπερβολικό περιθώριο ερμηνείας. Επίσης, όσον αφορά ε, τις στρεβλώσεις, θα πρέπει να έχουμε κατάλογο, όπως προτείνει ο κύριος Σίκου, αλλά θα πρέπει να είναι μη εξαντλητικός ο κατάλογος αυτός, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία ευελιξίας. Και όσον αφορά την ε, έκθεση, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται κάποιο είδους εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να είμαστε βέβαιοι έτσι ότι έχουμε μια καλή ανταλλαγή με τους διάφορους ενδιαφερομένους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Προύστ. Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον Σαλβατόρε Τσίκου, για τη δουλειά που έχει κάνει και κυρίως για την ποιότητα των τροπολογιών του. Και τον συγχαρώ επίσης γιατί δεν ήταν εύκολο να καταλήξει σε συμβιβαστική θέση όσον αφορά τον ορισμό των σημαντικών στρεβλώσεων κάτι που όλους μας απασχόλησε, ή πώς θα συμπεριληφθούν τα παλιά κριτήρια για την οικονομία της αγοράς, το οποίο νομίζω ότι με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία τα συμπεριλαμβάνει. Επίσης, είναι σημαντικό να το πούμε στην έκθεση και συνάδει με ακούσαμε μέχρι τώρα, ότι είναι σημαντικό να καθορίσουμε τον ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην εκπόνηση των εκθέσεων αυτών που προτείνονται. Θα διευκρινίσω στις επόμενες μέρες κάποια σημεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Και εδώ συμφωνώ με τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Μανουέλ Μορέλ, διότι πράγματι πρέπει να τις προστατεύσουμε. Ακριβώς εξαιτίας του μεγέθους τους, γιατί το μέγεθος παίζει ρόλο εδώ. Θα προσπαθήσω να καταλήξω σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Συμβαστικές δηλαδή από τη μια να προσφέρουμε στην Επιτροπή και στη βιομηχανία ε, να διαθέτει ευελιξία για να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους, αλλά από την άλλη μεριά, και το είπα και στην πρώτη ανάγνωση, να μην καταλήξουμε εδώ πέρα σε κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε πια να ελέγξουμε, που θα μας ξεφύγει εντελώ από τα χέρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω ότι θα μας δώσει κάποιες εγγύσεις για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για να εφαρμόσει τη νέα μεθοδολογία γιατί πρόκειται για τράπεζα δεδομένων, για μια παρακολούθηση που σημαίνει ότι χρειάζονται πόροι και ανθρώπινοι και οικονομικοί. Τι μέσα λοιπόν θα έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το, το μηχανισμό αυτό να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά και μάλιστα με τη νέα μεθοδολογία, τη, τον εξυγχρονισμό, αυτά πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτον, πρέπει να πετύχουμε μέγιστη αποτελεσματικότητα της νέας νομοθεσίας αντι-dumping με αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεύτερον, η συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ είναι ζωτική σημασίας. Οπότε, χαίρομαι για την πρόταση του εισηγητή, αλλά έχω δύο σχόλια. Πρώτον, πιστεύω όπως ήδη υπόθηκε από τους συναδέρφους ε, του σοσιαλιστές και το ECR, ότι το βάρος της απόδειξης να μην εμπίπτει στους, ε, να μην πέφτει στους ώμους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεύτερον, όταν μιλάμε για σημαντικές ε, στρεβλώσεις, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και τις στρεβλώσεις για κάθε τομέα παραγωγής. Και έχω και δύο ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα όσον αφορά το πάνελ του ΠΟΕ. Σε τι βαθμό μπορούμε να ελέγξουμε το πάνελ αυτό του ΠΟΕ και θα γίνεται με τη νέα νομοθεσία. Και έχω και μια ερώτηση προς τον εισηγητή λέτε στην έκθεσή σας, κάνετε τη σχέση με την νομοθεσία που ισχύει στι ΗΠΑ. Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερο πόσο μακριά θέλετε να πάτε, δηλαδή. Μιλήσατε για συγκριτικές μελέτες. Πώς ακριβώς το βλέπετε. Ευχαριστώ και τέλος ο κύριος Φερό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι μια έκθεση γεμάτη παγίδες. Ε, μιλάω εκ μέρους του Ματές Σαρβίνη, του σκιώδους εισηγητή της ομάδας μας που δεν μπορεί να είναι εδώ. Και ο συντονιστής της ομάδας επίσης. Η θέση του κύριου Τσίκου σίγουρα αποτελεί βελτίωση της νομοθετικής πρότασης, αλλά είναι προβληματική και με πολλά κενά. Πρέπει να δουλέψουμε βέβαια βάσει της πρότασης του εισηγητή για να καταλήξουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την προστασία των ε, ευρωπαϊκών βιομηχανιών και των μικρών και μεσών επιχειρήσεων γιατί η προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ μπορεί να μας εμποδίσει τελικά να έχουμε στη θέση μας μηχανισμούς για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας. Οι Κινέζοι είναι επιθετικοί πολλές φορές και μάλιστα εκτός οικονομίας της αγοράς. Έχω να προτείνω τρεις βελτιώσεις κύριε Τσίκου στην έκθεσή σας. Πρώτον, το βάρος της απόδοξης πρέπει να πέφτει στους ώμους των Κινέζων και ποτέ στους ώμους Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Δεύτερον, το κόστος της παραγωγής πρέπει να συμπληρωθεί για να εντοπίζονται καλύτερα οι παραβιάσεις και κίνδυνοι για τις βιομηχανίε μα. Και τρίτον, το να μιλάμε για σημαντικές τρευλώσει τη αγορά πρέπει να ε, καθορίζονται πολύ συγκεκριμένα. Προσοχή γιατί μπορεί να καταλήξει να είναι επικίνδυνη μια τέτοια διατύπωση έτσι όπως έχει τώρα. Αυτά λοιπόν τα τρία έχω να συμπληρώσω στην έκθεσή σας. Και δυστυχώς όπως πάντα τα προβλήματα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομοθετική πρόταση είναι αποδύναμη και λίγο αποτελεσματική. Και πολύ επιπόλαια. Για άλλη μια φορά δίνουμε τη δυνατότητα στους Κινέζους να χρησιμοποιούν πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς η Ευρώπη βρέθηκε μόνη της και χωρίς προστασία σε μια παγκόσμια αγορά χωρίς κανόνες. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα για μας τους Ευρωπαίους να αλλάξουμε την κατάσταση, γιατί η μεταφορά των επιχειρήσεων, η παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά ε, μας κάνει να μην μπορούμε να είμαστε όπως θα θέλαμε, αρκετά επιθετικοί δηλαδή και να υποστηρίζουμε τη βιομηχανία μας όπως θα θέλαμε. Πρέπει να βρούμε και συμμάχους όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες ή η Ιαπωνία, που έχουν δείξει ότι ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν για να αντιμετωπίσουν τον αθέμητο αντιγωνισμό. Ευχαριστούμε και η Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίκου για την ε, έκθεσή του. Και συμφωνώ με τον κύριο Μορέλη για τις τροπολογίες που θα προτείνει όσον αφορά τους παράγοντες ε, και τους κοινωνικούς και τους περιβαλλοντικούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις σημαντικές ε, στρεβλώσεις. Οι εκθέσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό στην νομοθεσία αυτή και όσον αφορά το βαρός της απόδειξης και όσον αφορά τις σημαντικές τρευλώσεις αυτές καθ' αυτές. Τώρα, ρωτάω την Επιτροπή. Έχουμε την απόδειξη ότι την έκθεση αυτή θα την έχουμε όταν θα ψηφίσουμε την νομοθεσία, γιατί μπορεί να συμφωνήσουμε επί της αρχής του να δουλεύουμε πάνω στην έκθεση που αποτελεί το κύριο στοιχείο της νομοθεσίας, αλλά θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ήδη μία έκθεση, κυρίως για την Κίνα, όταν θα ψηφίσουμε επί της νομοθεσίας αυτής. Αλλιώς δεν θα έχουμε την εγγύηση ότι το βάρος της απόδειξης δεν πέφτει στους ώμους της δικιάς μας βιομηχανίας. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρωτάω, έχει ήδη εκπονήσει μία στάνταρτ έκθεση σχετικά με την Κίνα, για παράδειγμα. Λοιπόν, μετά από την δική μου παρέμβαση θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά το Συμβούλιο. Πέντε λεπτά στον καθένα. Και σας παρακαλώ να επικεντρωθείτε στο ε, ε, ερώτημά μου και στα καυτά θέματα, διότι είχαμε μια γενική ανταλλαγή απόψεων, είχαμε και μια ακρόση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι... Υπόθηκε ότι κάποια μέλη του η Ρωσία, η Επιτροπή του Κόλπου, ε, το Καζακστάν, η Ινδονησία και άλλοι στήριξαν ε, το αίτημα της Κίνας ε, και είπαν ότι, υπάρχει, ότι η σημαντική στρέβλωση δεν έχει οριστεί πολύ σωστά. Λοιπόν, υπάρχει βάσιμος λόγος υποψίας ότι η πρότασή μας δεν ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Έχουμε την περίπτωση του βιοντίζελ με την Αργεντινή. Μπορούμε να υπερασπιστούμε την πρόταση αυτή και συμφωνώ με το ερώτημα του κ. Βαλένσα στο θέμα αυτό. Ή μήπω θα πρέπει να σκεφτούμε τις εκκρεμότητες ε, από το πρωτοκόλλο προσχώρησης διαφόρων χωρών. Ε, Κομισιόν πέντε λεπτά και μετά Συμβούλιο πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του και για την δέσμευσή του να ασχοληθεί με αυτό το πολύπλοκο θέμα εις βάθος. Επικροτούμε το γεγονός ότι η έκθεση διατηρεί τον πυρήνα και τη γενική προσέγγιση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά την ουδετερότητα του Συμβουλίου, το θέμα του ορισμού των ε, σοβαρών στρεβλώσεων και την ανάγκη να διατηρηθούν αποτελεσματικά μέσα άμυνας στο εμπόριο, παραμένοντας όμως ε, ευθυγραμμισμένοι με τις υποχρεώσεις ε, που επιβάλλει ο ΠΟΕ. Κάποιες από τις τροπολογίες που προτείνονται μας προκαλούν κάποιες, κάποιους ενδιασμούς όσον αφορά την νομιμότητα. Για παράδειγμα υπάρχει εδώ πέρα ένα στοιχείο αναδρομικότητας. Επίσης υπάρχει μια νομική προϋπόθεση με την οποία δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε και κάποια θέματα όσον αφορά την λειτουργικότητα αυτού του κανονισμού. Σημειώνω ότι εκφράστηκαν κάποιοι ενδιασμοί από διάφορους ευρωβουλευτές. Ε, ακούστηκαν και στο Συμβούλιο όταν το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση αυτή. Και είμαι βέβαιος ότι και ο συνάδελφος από την Προεδρία θα το πει αυτό. Το Συμβούλιο κατάφερε να καταλήξει σε καλή λύση που ε, έγινε απόλυτα αποδεκτή ε, με ομοφωνία. Το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό επικροτούμε και την ε, δέσμευση και την αφοσίωση του εισηγητή. Τελικά, σημαντικό για την ε, βιομηχανία είναι η ασφάλεια δικαίου. Και το να μην ισχύει ένας τέτοιος κανονισμός δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια. Θα αναφερθώ σε κάποιες από τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Το θέμα του βάρους της απόδειξης πιστεύουμε ήδη έχει λυθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όπως και στον συμβιβασμό του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει εάν υπάρχει κάποιο σοβαρή στρέβλωση. Δεν το αποφασίζει αυτό κάποιος άλλος. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίσει μια τέτοια στρέβλωση, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την εναλλακτική μεθοδολογία και αν διαφωνεί κάποιος εξαγωγέας, ε, θα πρέπει αυτός να αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λάθος. Όσον αφορά τον κατάλογο στρεβλώσεων, σημειώνουμε ότι καταρχάς ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη είναι ανοιχτός ο κατάλογος αυτός, μπορούμε να προσθέσουμε όσες προτάσεις θέλουμε στον κατάλογο αυτόν, αλλά θα πρέπει πρώτον να φροντίσουμε να μην ξεπεράσουμε την γραμμή της συμμόρφωσης με τον ΠΟΕ και να φροντίσουμε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να διαπιστώσει στρέβλωση με βάση τα κριτήρια αυτά, ώστε η νέα εναλλακτική μεθοδολογία να μπορεί να εφαρμοστεί. Όσον αφορά τις κυρώσεις για μη συνεργασία, ε, σημειώνω την παρατήρηση του κυρίου Μαρέλ, ε, τα άρθρα 18 και 28 αντίστοιχα των κανονισμών anti-dumping ε, και για τις επιδοτήσεις αποτελούν βάση για συνεργασία και όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα ισχύοντα μέτρα έχουμε πολλά μέτρα τα οποία ισχύουν για τομείς όπου συμμετέχει μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά την συμμόρφωση με τον ΠΟΕ, να είμαστε απόλυτα σαφείς. Θεωρούμε ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα μπορούσε οποιοδήποτε μέλος του ΠΟΕ να επιτεθεί σε μας ε, για νομοθεσία που δεν ισχύει ακόμα. Σίγουρα είμαστε διατεθειμένοι να υπερασπιστούμε στο βαθμό που μπορούμε και την ισχύουσα νομοθεσία. Όπως είπε όμως ο κύριος Σίκου, σημαντικό είναι να συμμορφωνόμαστε με τον ΠΟΕ, αλλά να παραμένουμε και αποτελεσματικοί. Όσον αφορά τον ε, ορισμό των εκθέσεων, η βιομηχανία θα έχει πολλές ευκαιρίες να σχολιάσει τις εκθέσεις αυτές ε, κατά τη διάρκεια των ερευνών και νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να εξαλείψουμε οποιοδήποτε άχθος για τη βιομηχανία ή να ε, δώσουμε στη βιομηχανία τη δυνατότητα να αναπτύξει επιχειρήματα για το γιατί υπάρχουν ε, στρεβλώσεις. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι η αρχή του προϋπολογισμού ε, δεσμεύεται όμως να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του ε, κανονισμού αυτού, γι' αυτό θα διαθέσουμε ε, τους απαραίτητους πόρους. Επίσης, στην κυρία Ρένα να πω ότι έχουμε ε, σχεδιάσει την εκπόνηση μια έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια έκθεση όσο γίνεται πιο σύντομα. Επίση, η κυβέρνηση των Ηνωμένων έχει ξεκινήσει αναθεώρηση, επικαιροποίηση του ισχύ, της ε, παρούσας έκθεσης και θα τα μεταφέρω όλα αυτά στην Επίτροπο Μάλμστρομ για να δούμε πώς μπορούμε να ε, παράσουμε περαιτέρω ε, εγγυήσεις και διασφαλίσεις στο Κοινοβούλιο πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο υιοθέτησε ε, σχετικά σύντομα την διαπραγματευτική εντολή, κάτι που μας εξέπληξε. Ιδιαίτερα σε σύγκριση με, το, με τη δέσμη μέτρων για τον εξυγχρονισμό, κάτι που σε τρία χρόνια. Δίνω λοιπόν το λόγο στον πρόεδρο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το εμπόριο. Από την Μαλτέζικη Προεδρία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το σχέδιο του εισηγητή και τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα ε, αντιστοιχούν στις ίδιες ανησυχίες που έχουμε και στο Συμβούλιο. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με την Κομισιόν και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συναδέλφο από την Κομισιόν. Συμφωνούμε γενικά και θεωρούμε ότι η συμμόρφωση με τον ΠΟΕ αποτελεί το κλειδί της πρότασης αυτής. Έχουμε ήδη πράγματι υιοθετήσει τη θέση μας από χθε στην Κορεπέρ. Όπως λέτε κύριε Λάγκε, πρόκειται για μία ε, σπάνια κατάσταση. Και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και τους υπόλοιπους, διότι αυτό κατέστη δυνατόν, διότι το Συμβούλιο ε, ήταν ανοιχτό να ακούσει όλα τα σχόλια του Κοινοβουλίου ε, και να επιταχύνει ε, τις διαδικασίες ε, εμπορικής άμυνας. Και αυτό και επιτύχαμε. Αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας Προεδρίας. Ο Συμβούλιο μας απασχολεί λόγω του πολιτικού και νομικού πλαισίου η αναγκαιότητα να δράσουμε γρήγορα ω ε, συνολική Ευρωπαϊκή Ένωση με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Συμβούλιο κατάφερε σε λιγότερο από έξι μήνε μετά από την ε, δημοσιοποίηση τη πρόταση αυτή να καταλήξει σε μια ενιαία θέση που διατηρεί το πνεύμα της πρότασης της Κομισιόν ενώ ενισχύει με νομικά ε, υγιή τρόπο τις διατάξεις διασφάλισης προσπελάσιμου και παρεμφερούς επίπεδου προστασίας ε, για τους Ευρωπαίους βιομηχανούς. Το Συμβούλιο είναι της άποψη ότι το τελικό προϊόν της νομοθετικής διαδικασίας πρέπει να είναι ε, συμμορφούμενο με τον ΠΟΕ οπωσδήποτε και ότι πρέπει να ανταποκρίνεται στις ε, ε, ανάγκες της βιομηχανίας κυρίως όσον αφορά τις εκθέσεις. Το Συμβούλιο επισημοποίησε το, την εσωτερική του εντολή για τι διαπραγματεύσει και είναι έτοιμο να ξεκινήσει τι διοργανικέ συζητήσει μόλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, καθορίσει την τελική του θέση. Λόγω τη ευαίσθητη φύση του θέματος αυτού θεωρούμε ότι η ευθυγράμμιση και η ενότητα εντός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τέλος, η Προεδρία θα ήθελε να ενθαρρύνει την Επιτροπή ΕΝΤΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ όφελο όλων των ενδιαφερομένων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσουν πολύ γρήγορα μια θέση. Φιλοδοξία μα είναι να ολοκληρώσουμε μαζί ω νομοθέτε την νομοθετική διαδικασία και να τεθεί η νέα νομοθεσία σε ισχύ πριν το καλοκαίρι, ώστε να διασφαλιστεί άμεση συνέχιση της προστασίας κατά του ντάμπινγκ για τη βιομηχανία μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών ε, αμυντικών ε, μέσων άμυνας του εμπορίου για το άμεσο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σίκα, ε, θέλατε να κλείσετε κύριε Τσίκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω ειδικότερα όλους τους συναδέλφους ε, που παρενέβησαν. Πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά θα χρειαστούν επιπλέον αλλαγές, προσθήκες, προτάσεις. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, μεταξύ άλλων, ε, για όσα, με όσα υπόθηκαν για τα κοινωνικά θέματα, πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα και από νομική άποψη Συμφωνώ και με κάποιες παρατηρήσεις ορισμένων συναδέλφων, ε, στις οποίες θέλω να επανέλθω εν συντομία. Νομίζω ότι κατέστησα σαφέ όσον αφορά τα θέματα της, ο βάρος της απόδειξης, τις τροπολογίες μου, το βάρος της απόδειξης ε, ορίζεται από την έκθεση της Κομισιόν για ένα συγκεκριμένο τομέα, για μια συγκεκριμένη χώρα διότι εκεί θα ε, προσδιορίζεται κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια που οδηγούν σε σημαντικές τρευλώσεις. Η συγκριτική ανάλυση με το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη συμπεριληφθεί στο σύστημα αυτό, διότι η έκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών ουδέποτε σε διάκριση Κίνας ε, ως οικονομίας αγοράς ή όχι. Απλά ε, διαπιστώνει κατά πόσο πληρούνται οι συνθήκε οι οποίε πραγματοποιούν τη διάκριση μεταξύ οικονομία αγορά ή όχι χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη χώρα διότι αυτό είναι το νομικό σημείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς υπερασπισή μα. Το βάρος λοιπόν τη απόδειξης διαφυλάσσει τη θέση τη δική μα βιομηχανία, απόλυτα διότι μόνο μία χώρα εξαγωγική αφού δοθεί το βάρος της απόδειξης ε, στην εκθέση της Κομισιόν μπορεί να δώσει τα δικά του αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει ότι δεν βρίσκεται στη θέση στην οποία τον θέτει, τη θέτει η έκθεση. Να δώσω το παράδειγμα ενός κριτηρίου γιατί άκουσα κάποιες αξιολογήσεις ε, που κατ' εμέ τεχνικά δεν έχουν νόημα. Όταν μιλάμε για το δίκαιο περιχροκοπίας μιας χώρας, το δίκαιο αυτό δείχνει αν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προστατεύει με χρηματοδοτήσεις, με πρόσβαση χρηματοδοτήσεις, με ε, συγκεκριμένους πόρους, διότι στις ευρωπαϊκές χώρες ε, χρεοκοπεί μια εταιρεία διότι υπάρχει ελεύθερη πρωτοβουλία, διότι μια επιχείρηση ε, επενδύει στον εαυτό της. Εάν δεν χρεοκοπήσει μια εταιρεία, το, το, το ε, εταιρικό δίκαιο ε, είναι διαφανές όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εξετάζω εγώ. Θεωρώ ότι όλα τα σχόλια που ακούσαμε ήταν σημαντικά και πολύ χρήσιμα για να ε, τελειοποιήσουμε την πρότασή μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σκληρή σας δουλειά. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 18η Μαΐου. Σχετικά σύντομα δηλαδή. 12 η ώρα το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή στις 20 Ιουνίου. Και αυτό αρκετά σύντομα δηλαδή, ώστε να ε, λειτουργούμε παράλληλα με το Συμβούλιο που επίσης κινήθηκε πολύ γρήγορα επί το αρχείο αυτού. Προτείνω να αναβάλουμε τα στοιχεία 22 και 23 για μετά την ψηφοφορία. Οπότε ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. And the first item is... Το πρώτο θέμα, λοιπόν, για το οποίο θα ψηφίσουμε είναι το σημείο 24. Το πρώτο θέμα που θα ψηφίσουμε είναι το σημείο 24. Διάθεση προϊόντων λίπανσης. Πρωτού προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε αν έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί σας. Έναρξη λοιπόν της δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Haben Sie alle abgestimmt? όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Όλα εντάξει. Και εσάς παρακαλώ. Ησυχία. Μπορείτε ή να σοπάσετε ή να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Δύο επιλογές έχετε. Προχωράμε λοιπόν στο σημείο 24. Και ψηφίζουμε. Συζητήσαμε με τον εισηγητή, δυστυχώς. Κάποιες τροπολογίες ε, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και δεν θα μπορέσουμε να τις ψηφίσουμε εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν από τη συμβαστική ψηφοφορία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, Επαλήθευση. Τροπολογία 10. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. ist geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία πάνω στην έκθεση έναρξης ψηφοφορίας. Und Abstimmung ist Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, συγχαρητήρια κύριε Βαλέσα. Προχωράμε στο σημείο 25. Um, das ist der που έχει να κάνει με την προσχώρηση στην Επιτροπή ε, Βαμβακιού, έναρξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Σημείο 26. Πρώτο ψηφίσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Ρούας έχει αποσύρει τις ε, τροπολογίες 1, 2, 4 και 5. 1, 2, 4 και 5. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Μολδαβία. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αφέτ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 και 15 της ΑΦΕΤ είναι πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 16 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της ΑΦΕΤ λέει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 της αφέτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της αφέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαέξι, ωστόσο, όχι ολόκληρη, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Έναξη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ο εισηγητής θέλει να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις. Κύριε Μωυσά, θα ψηφίσουμε πάνω και σε αυτό το θέμα λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ. Μάλλον όχι, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας για το εάν θέλουμε να ξεκινήσουμε σε ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις. Η λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Σημείο 27. Προσωρινά αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την Ουκρανία. Επίσης έκθεση του κυρίου Βαλέσα. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ε, συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, συμβαστική τροπολογία 9, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Änderungsantrag 22. Ε, ε, τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι την τροπολογία 25, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας. Τροπολογία 3. Συγγνώμη, καταπίπτει. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ξέχασα την ε, ε, τροπολογία 7 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Θερμά συγχαρητήρια. Και φτάνουμε στην προφορική ερώτηση για τον Μπαγκλαντές. Μία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Und Abstimmung ist geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας. Σχεδόν ομόφωνα ψηφίστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και επανερχόμαστε στο σημείο 22. Κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ε, των τριμερών διαλόγων. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται τριμερής διάλογος ε, για τον εξυγχρονισμό των ε, εργαλείων ε, προστασίας του εμπορίου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τριμερή διάλογο για κάποια τεχνικά ζητήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εάν αποχωρείτε από την αίθουσα, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα. Για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Πραγματοποιήθηκε σε διάλογος για τα τεχνικά ζητήματα του εξυγχρονισμού. Ήταν επικοδομητική συνάντηση αυτή. Βρήκαμε κάποιες, καταλήξαμε σε κάποιους συμβιβασμούς με το Συμβούλιο. Τα αποφασιστική σημασίας πολιτικά ζητήματα, για παράδειγμα η λεγόμενη ρήτρα shipping ναυτιλίας, το πόσο πριν θα πρέπει να ε, γίνεται η ενημέρωση ή Ε, ο κανόνας ε, σχετικά με τους χαμηλότερους δυνατούς ε, δεσμούς. Αυτά τα ζητήματα δεν συζητήθηκαν, θα συζητηθούν κατά τον επόμενο τριμερή διάλογο που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Ερωτήσεις υπάρχουν, όχι. Προχωράμε στο σημείο 23, παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων. Είχαμε μία για τη Ρωσία στις 23 Μαρτίου. που είχε να κάνει με τις, ρωσικές με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Ρωσία. Ο κύριος Στάκουλα δεν είναι παρόν, άρα δεν μπορεί να συμπληρώσει τίποτα. Κατόπιν ε, είχαμε συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης Mercosur. Ε, ο κύριος Αρφράγκα είναι παρόν, μπορεί να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, γιατί πρέπει να φύγω τρέχοντας για το αεροδρόμιο. Η ομάδα ελέγχου συνεδρίασε όντω την προηγούμενη εβδομάδα με τον επικεφαλή των διαπραγματεύσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν όλοι περίπου ισχυώδει εισηγητέ και είναι 27η, 27ος γύρος αυτής της μακράς ε, συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μερκοσούρ. Αυτή, αυτός ο τελευταίος γύρος έγινε στο Πένος Άιρες υπό την Αργεντινή Προεδρία της Μερκοσούρ και σημειώθηκε πρόοδος στα 15 κεφάλαια που είναι ανοιχτά τώρα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τα εμπόδια βέβαια παραμένουν στα πιο ευαίσθητα σημεία που είναι το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και σε άλλα ευαίσθητα κεφάλαια όπως είναι οι δημόσιες αγορές υπήρξε κάποια πρόοδος. Η επικεφαλής από τη διαπραγματευτική ομάδα της Κομισιόν μας είπε ότι θέλει να εποφεληθεί από αυτή την εποχή που οι τέσσερις χώρες της Μερκοσούρ είναι στο ίδιο περίπου κλίμα. Το ίδιο ισχύει και με την αλλαγή στις προτεραιότητες. Μετά από την εκλογή του Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείες είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προσπαθήσει να κλείσει την διαπραγμάτευση αυτή προς τα τέλη της χρονιάς. Όμως παραμένουν κάποιες δυσκολίες. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει με στόχο να κλείσει η διαπραγμάτευση στα τέλη της χρονιάς. Όμως το φθινόπωρο δεν ξέρω αν θα υπάρξει πολλή κίνηση. Αυτή είναι η πορεία. Δηλαδή κάποια λογική πρόοδος, αλλά παραμένουν ευαίσθητα ζητήματα που όπως ξέρουν οι συνάδελφοι είναι τα γεωργικά προϊόντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπηρεσίες για τους εταίρους μας από την ε, Μερκοσούρ. Αυτά πρέπει να λυθούν ακόμα. Ο ρυθμός της διαπραγμάτευσης βαίνει καλός, είναι έντονος. Και όπως μας εξήγησε η επικεφαλής, επανέλαβε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσπαθήσει να υποφεληθεί από την ευκαιρία που δίνεται βάση της συγκυρίας για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε στα τέλη της χρονιάς. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Στο μεταξύ, πρέπει να υπάρξει νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευαίσθητα σημεία και ενδεχομένω και απόφαση των Υπουργών Εμπορίου ενδεχομένως. Αυτά γενικά κάπως, Πρόεδρε. Τα πιο σημαντικά στοιχεία από τις πληροφορίες που έχουμε από την επικεφαλής ε, των διαπραγματεύσεων της ε, Επιτροπής είναι ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτά ακούγονται όλα πολύ θετικά. Πολύ αισιόδοξα διαπραγματεύσεις ε, στη Μερκοσούρ ε, ε, γίνονται εδώ και 10 χρόνια. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία λοιπόν. Χιλή. Χθε συζητήσαμε το θέμα αυτό, χθε ει βάθο εδώ στην Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε. Κατόπιν έχουμε ASEAN και VSP. Κοινή συνάντηση στι 27 Απριλίου. David Martin. Δεν μπορούμε λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό. Και τώρα έχουμε την παρακολούθηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ε, και της Φιλιππίνες. Αυτό θα πρέπει να το αναβάλουμε. Και τέλος έχουμε την Ιαπωνία στις 3 Μαΐου. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Σίλβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Καλό θα ήταν να πιστήσω την προσοχή σας στο ότι έχουμε μια ομάδα παρακολούθησης ε, για την Ιαπωνία ε, η οποία συνήλθε χθε. Εκεί είχαμε την ενημέρωση του κυρίου διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κυρίου Πετριτσάνη, για τον ε, προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα την εβδομάδα της 3ης Απριλίου οι διαπραγματεύσει από ιαπωνικής πλευράς τώρα διευθύνονται από ένα νέο διαπραγματευτή, τον τέταρτο, τον ε, πρέσβη Σουζούκη. Ήταν δημόσιος αυτός ο γύρος, ε, το ίδιο και πολλές ευρωπαϊκές προτάσεις και ε, συμπεριλαμβανόμενες της ρυθμιστικής συνεργασίας. Κάτι που εμείς καλωσορίζουμε. Οι διαπραγματευτές έχουν προγραμματίσει τακτικές και εντατικές συναντήσεις για τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει μια συνάντηση ήδη μέσα Μαΐου. Να υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο ο, κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Χάμπεϊ με τον κύριο Τάσκη και Γιούνκερ ε, επανεπιβεβαιώσαν τη δέσμευσή τους για μια επί της αρχής συμφωνία των νωρίτερων δυνατών. Και τέλος, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή σημειώνεται σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς. Ο κύριος διαπραγματευτής χρησιμοποίησε τα μαγικά λόγια. Μπαίνουμε στην τελική φάση. Ας δούμε αν είναι αλήθεια πολλά κεφάλαια όπως η βιώσιμη ε, ανάπτυξη ε, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί αλλά κάποια σημαντικά ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ε, τα γεωργικά προϊόντα, οι δημόσιες συμβάσεις και το σύστημα επίλυσης επενδυτικών διαφορών και η συμφωνία θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί καλό αποτέλεσμα για όλα αυτά τα ζητήματα κλειδιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε την Ιαπωνία στην Επιτροπή μας ε, ε, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Καλά ακούγονται τα πράγματα. Ε, οικονομικά φυσικά η Ιαπωνία είναι πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Εδώ ολοκληρώνεται τα διάφορα, το σημείο αυτό και περνάμε στο 29 στην ακρόασή μας και τη συζήτηση περί κανόνων καταγωγής. Οι κανόνες καταγωγής είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στις ε, εμπορικές σχέσεις, διότι έτσι διασφαλίζεται, ρυθμίζεται η δυνατότητα των διαφόρων χωρών ε, να συμμετάσχουν στο διεθνές εμπόριο. Εν τω μεταξύ, όλο και λιγότερο ισχύει ένα προϊόν να παράγεται κατά 100% σε μία χώρα. Γι' αυτό το θέμα των κανόνων καταγωγής είναι πολύ κεντρικό στις εμπορικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, με τον Καναδά, στο πλαίσιο τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, διαπραγματευτήκαμε πολύ εντατικά ε, πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, ένα καναδικό αυτοκίνητο πότε είναι καναδικό και πότε είναι αμερικανικό. Ή, για παράδειγμα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ιορδανία να εντάξει τους ε, πρόσφυγες ε, στην ε, διαδικασία παραγωγής και μήπως μπορούμε να χαλαρώσουμε τους κανόνες και τι ισχύει για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και πώς μπορούμε να φέρουμε τα προϊόντα της Ιορδανίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Πολύ κεντρικό θέμα στην εμπορική πολιτική λοιπόν και γι' αυτό Χαίρομαι που μπορούμε τώρα να το συζητήσουμε. Στον πρώτο γύρο μας, στον πρώτο γύρο της συζήτησης θα ακούσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα του κυρίου Χέντριξ που είναι αρμόδιος για τους κανόνες ε, καταγωγής από την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ε, και θα ακούσουμε και τον κύριο Ιγνάθιο Ιρουαριγάς Διές, ε, που είναι τμήματάρχη στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Κύριε Χέντριξ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Uh, Ζητώ συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την παρουσίαση, με τις διαφάνειες προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Albert Χέντριξ και είμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις και για την διαχείριση των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Διαπραγματεύτηκα την ΣΥΤΑ, TTIP, μέχρι που σταματήσαμε και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε και τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Πρώτα απ' όλα, μπράβο που δείχνετε ενδιαφέρον για ένα τόσο τεχνικό θέμα όπως είναι αυτοί οι λεγόμενοι κανόνες καταγωγής για το εμπόριο αγαθών. Ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μας το θέμα αυτό και θα προσπαθήσω στην παρουσίασή μου να σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. καθορίζουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει το καθεστώς ε, το δασμολογικό ευνοούμενης χώρας. τα ωφέλη περιορίζονται σε προϊόντα τα οποία παράγονται σε συγκεκριμένες επικράτειες και από συγκεκριμένους εμπορικούς εταίρους. Η καταγωγή αυτή είναι λιγάκι σαν να μιλάμε για την υπηκότητα του προϊόντος που καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων φυσικών παραδοσιακών δεσμών με την επικράτεια από όπου παράγονται. Βέβαια, περνάμε από διαπραγματεύσεις για να αποφασίσουμε την πρόσβαση των προϊόντων αυτών στις αγορές μας και να βάλουμε υπόψη διάφορους παράγοντες. Είναι περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα βέβαια οι διάφοροι παράγοντες και όχι πολιτικοί για να αποφασίσουμε και ποιος αποφελείται και ποιος δεν αποφελείται από αυτούς τους κανόνες καταγωγής. Αυτά στην θεωρία βέβαια, γιατί θα σας εξηγήσουμε την εμπορική πολιτική που απορρέει από τους κανόνες αυτούς καταγωγής όπως λέγονται. Υπάρχουν οι μη προτιμησιακοί, πρώτα απ' όλα, που είναι μια άλλη κατηγορία και που εφαρμόζονται για διαφορετικούς λόγους από ότι οι προτιμησιακοί δασμοί κυρίως για λόγους εμπορικής προστασίας, αντι-dumping, ε, κατά των επιδοτήσεων, ποσοστώσεις, ρήτρες ασφάλειας. Και υπάρχουν κάποια κοινά αλλά και διαφορές μεταξύ των ε, προτιμησιακών κανόνων και των μη προτιμησιακών κανόνων. που εφαρμόζονται στις διάφορες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω πρώτα κάποιες βασικές αρχές της προτιμησιακής προέλευσης. Και έχω εδώ πέρα αυτήν την ε, παρουσίαση PowerPoint. Τρεις κατηγορίες, κύριε, υπάρχουν τέτοιων ε, κανόνων καταγωγής. Ανάλογα Βέβαια, συχνά μιλάμε για κατηγορία νόμου καταγωγής, εκεί που αναφέρονται γενικές διατάξεις, προκειμένου ένα προϊόν να αποκτήσει το καθεστώς αυτό. Και υπάρχει και ένα τμήμα Β, που περιλαμβάνει τις διαδικαστικές διατάξεις, πώς ε, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ή να αποδείξει ότι μπορεί να υποφεληθεί από μια τέτοια προτιμησιακή μεταχείριση. Και το τρίτο στοιχείο είναι οι ειδικοί κανόνες προϊόντων. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επεκταθώ λιγάκι τώρα σε αυτά τα τρία στοιχεία. Τμήμα Α. Γενικές διατάξεις. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια απλή διάκριση, πολύ βασική όμως. Πώς δηλαδή αποφασίζεται το ποια είναι η καταγωγή των προϊόντων. Ένα προϊόν αποκτά αυτό το χαρακτηρισμό καταγωγής είτε πλήρως είτε καλαμπόκι που γίνεται συγκομιδή ή που ψαρεύουμε τα ψάρια ή προϊόντα καλύπτουν μερικώς μόνο τα κριτήρια αυτά καταγωγής. Και υπάρχουν ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις για πολλά προϊόντα που έχουν να κάνουν με τους ειδικούς κανόνες προϊόντος. Αν δούμε τώρα την συνολική αλυσίδα, θα λέγαμε ότι η συζήτηση αυτή επικεντρώνεται κυρίως στους ειδικούς κανόνες προϊόντος. Βέβαια και άλλες διατάξεις παίζουν ρόλο, πως είναι η συσσόρευση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος, προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένα προϊόν παράγεται από υλικά που προέρχονται επίσης από το ίδιο μέρος. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες στις γενικές διατάξεις που έχουν να κάνουν και μία αρνητική δοκιμή. Αν δηλαδή ανακατέψεις προϊόντα υλικά, ποτέ δεν θα καλύψει τους ε, κανόνες αυτούς ε, καταγωγής ένα προϊόν αν δεν περάσει τη δοκιμή αυτή. Έχει να κάνει με την αρχή της εδαφικότητας αυτό Κάπου 15 με 16 διατάξεις υπάρχουν για αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στις γενικές διατάξεις. Περνάμε τώρα κάπως σύντομα στις διαδικαστικές απαιτήσεις που έχουν αναπτυχθεί τις εξυγχρονίζουμε αυτή την εποχή, γι' αυτό και θα επανέλθω αργότερα στην παρουσίασή μου σε αυτές τις απαιτήσει. Και έρχομαι τώρα στους ειδικού κανόνες προϊόντος. Είπα ότι υπάρχουν τριών ειδών κανόνες. Για τους ειδικού κανόνες επίσης υπάρχουν τριών ειδών. Υπάρχει το πώς αποφασίζεται η καταγωγή ενός προϊόντος και έχει να κάνει με την ανώτερη αξία του υλικού που εισάγεται. Και υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσει για την αξία του υλικού αυτού που πρέπει να είναι τοπικό σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Αλλιώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι καταγωγή από τη συγκεκριμένη χώρα. Το δεύτερο κριτήριο στους ειδικού κανόνες είναι η αλλαγή στο δασμό, δηλαδή τα υλικά που σάγονται πρέπει να τυχαίνουν τέτοιας ε, διαδικασίας ε, παραγωγής που να μην θεωρείται ότι προέρχονται τελικά από διαφορετική χώρα. Και τέλος υπάρχουν και κάποιες ειδικέ απαιτήσει επεξεργασίας του προϊόντος. Για τα ρούχα, για παράδειγμα, οι απαιτήσει επεξεργασίας είναι τέτοιες που το υλικό πρέπει να έχει περάσει από τη διαδικασία κατασκευής στη συγκεκριμένη χώρα, ακόμα και το να έχει γναθεί εκεί. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με την αξία ή με τους δασμούς. Να πω και κάτι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις διαπραγματεύσεις για τους ειδικού κανόνες προϊόντος και καταγωγής. Και αυτό παγκοσμίω βέβαια, όχι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο ε, ασχολούμαστε με διαπραγματεύσει περισσότερο από ποτέ. Και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή στις ε, αξίες, είτε διμερός, είτε περιφερειακός. Επίσης έχουμε πολλές εμπορικές συμφωνίες. Έχουμε επίσης τις επιπτώσεις του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλές αλυσίδες αξίας των προϊόντων και σε διμερές αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο με τέτοιες συμφωνίες. εξαιτία της αλλαγής στην διαδικασία παραγωγής. Και επίσης, αλλά αυτό έχει σχέση με την πολυπλοκότητα αυτού που ονομάζουμε αλυσίδα αξίας είναι ότι οι διάφορες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μεταξύ τους είναι αλληλένδετες μερικές φορές. Οπότε υπάρχει μια συσσόρευση. Στην ΣΥΤΑ, για παράδειγμα, ή στη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη ή την Ιαπωνία που συζητάμε αυτή την εποχή και με το Βιετνάμ επίσης. Συζητάμε το θέμα της ισόρευσης και στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με την Ιαπωνία. Και τέλος υπάρχει αντιπαράθεση διαφορετικών παραδόσεων στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε και διαχειριζόμαστε την ε, προτιμησιακή καταγωγή. Βέβαια και οι εταίροι έχουν αναπτύξει το δικό τους μοντέλο, οπότε οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε τώρα είναι περισσότερο αντιπαράθεση διαφορετικών μοντέλων που έχουν αναπτύξει τα διαπραγματευόμενα μέρη. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τους τρεις πυλώνες για την ανάπτυξη νέων κανόνων. Πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, με περίπλοκες διαπραγματεύσεις, οπότε καλώς θα ήταν να δει κανεί πώς αναπτύσσονται οι νέοι κανόνες και να τους χωρίσουμε σε τρεις πυλώνες. Πρώτα απ' όλα θέλουμε πιο απλού κανόνες για να καθορίζουμε πιο απλά την προτιμησιακή καταγωγή και τα προγράμματα συσσόρευσης. Σημασία έχει επίσης η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, προκειμένου να λειτουργούμε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Εδώ επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην επανεξιολόγηση, γιατί θέλουμε, όπως είπα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικαστικών απαιτήσεων. Οπότε εδώ γίνονται συζητήσεις για να καθοριστούν οι ευθύνες που έχουν οικονομικοί φορείς και οι δημόσιες αρχές για να καθοριστεί ένα καθεστώς ελέγχου της προτιμησιακής καταγωγής. Άρα χρειάζεται μια παλήθευση, ένας έλεγχος από αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι χώρες που εξάγουν με πιστοποιητικό που εκδίδεται σε αυτές ακριβώς τις χώρες. Αυτή είναι μια διαδικασία που ίσως δεν έχει αρκετή διαφάνεια. Αποτέλεσμα αυτού Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει μια διαδικασία συνδέοντας τρεις αρχές. Η πρώτη αρχή είναι αρχή της αυτοπιστοποίησης από τους εξαγωγείς και αυτό με εμπορικά έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται ε, από τους εμπορικούς εταίρους. Αυτό βέβαια προβλέπει συνεργασία όσον αφορά την επαλήθευση της καταγωγής και υπάρχει και η αρχή της άρνησης της καταγωγής που μπορεί να γίνει αν τελικά φαίνεται στον εισαγωγέ ότι τα προϊόντα αυτά δεν προέρχονται όντως από την χώρα καταγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θέλει να ευνοήσει την αρχή αυτή της αυτοπιστοποίησης. Βέβαια υπάρχουν σημερινές συμφωνίες που επιτρέπουν στις κυβερνητικές αρχές να εκδίδουν τέτοια πιστοποιητικά. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαμε, υπάρχουν δυνατότητες για κυβερνητικές πιστοποίησεις που αναφέρουν την καταγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Για τις εξαγωγές προχωρούμε σε δηλώσεις καταγωγής. Απαιτούμε από τον εξαγωγέα να είναι καταγραμμένο σε μια βάση δεδομένων, μια απλή καταγραφή σε ένα μητρό αυτό φτάνει. Και δεν χρειάζεται έτσι πια, όπως ισχύει τώρα, να υπάρχει πρώτα έγκριση των δηλώσεων καταγωγής από τις αρχές που εξάγουν. Απομακρυνόμαστε δηλαδή από ένα σύστημα αδειοδότησης των εξαγωγών. Επίσης, όσον αφορά την επαλήθευση. Αυτό ήταν ο πρώτος πυλώνας. Έτσι. Περνάμε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Ο δεύτερος πυλώνας θα ήταν, όπως είπα, η αρχή της ανάγκης διοικητικής συνεργασίας για την επαλήθευση της καταγωγής. Αυτό είναι θέμα του χαρακτηρισμού καταγωγής. Πριν υπάρχει αίτηση για προτιμησιακή μεταχείριση οι αρχές που εισάγουν μπορούν να κάνουν τις δικές τους έρευνες. Ρωτώντας τον εξαγωγέ, τον παραγωγό και τις αρχές των εξαγωγικών χωρών. Δεν έχουμε προβλέψει απευθείας επαφή ανάμεσα στις αρχές που εισάγουν και τις εξαγωγικές αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διατηρείται το απόρριτο. Και συνήθως οι εξαγωγείς δεν θέλουν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αρχών που εισάγουν σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Το τρίτο στοιχείο είναι το θέμα της άρνησης. Προχωρούμε σε άρνηση της ε, προτιμησιακής μεταχείρισης βάσει της αξιολόγησης του εισαγωγέα, της πλευράς που εισάγει. Βάσει των δηλώσεων που έχει κάνει η εξαγωγική πλευρά. Οπότε πέφτει το βάρος στην πλευρά που εισάγει. Και έρχομαι και σε άλλη μια διαφάνεια που έχει να κάνει με το ασφαλές περιβάλλον. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί οι κανόνες προτιμησιακής μεταχείρισης ε, ισχύουν για την κάθε πλευρά χωριστά. Βέβαια υπάρχει μια κοινή διαχείριση που έχει να κάνει μόνο με την επαλήθευση της προέλευσης, με αμοιβαία διοικητική αρρωγή σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια έρευνα και κάποιες ειδικές επιτροπές που ελέγχουν τους κανόνες καταγωγής. Μερικές φορές προβλέπουμε κοινέ κατευθυντήριες γραμμές σε επεξηγηματικά σημειώματα μεταξύ των δύο πλευρών. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αναπτύξει τα προληπτικά μέτρα που πρόκειται επίσης για ανακοινώσεις που κάνουμε προς τους εισαγωγείς, σημειώματα, στην περίπτωση που υπάρχει κάποια απάτη, αλλά συνεισφέρουμε επίσης και στην οικοδόμηση ικανοτήτων στις άλλες πλευρές, αναπτύσσοντας ελεγκτικές δράσεις, αφού αρχίσουν, αρχίσει να ισχύει το καθεστώς αυτό της προτιμησιακής αντιμετώπισης. Και έτσι φτάνω στο τέλος της παρουσίασής μου και ελπίζω έτσι να σας έδειξα ποιες είναι οι βασικές αρχές για να καθοριστεί η καταγωγή ενός προϊόντος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χέντριξ. Παρακαλώ. Thank you, Chairman, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Επιτρέψτε μου να εμφανίσω τις διαφάνειες στην οθόνη. Ουσιαστικά δύο είναι οι περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι σημαντικοί οι κανονές καταγωγής δύο ε, τύπους εμπορίου που θέλουμε να απλουστεύσουμε υποπροτιμησιακό καθεστώς ε, και ε, όπου γίνεται διάκριση μεταξύ προϊόντων μιας χώρας και μιας άλλης και των περιπτώσεων όπου ισχύει η αρχή του πλέον ευνοούμενου κράτους που είναι αρχή του ΠΟΕ όπως γνωρίζουμε και στις δύο περιπτώσεις ε, λειτουργούν διαφορετικά οι κανόνες καταγωγής. Στην πρώτη περίπτωση όπου έχουμε την εφαρμογή της αρχής ε, του ΠΟΕ για το πλέον ευνοούμενο κράτος δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία οι κανόνες καταγωγής σε, αυτή την περίπτωση. Το υπογραμμίζω περιορίζονται στατιστικά. Όταν λοιπόν εφαρμόζονται οι κανόνες MFN, όταν στο πλαίσιο μιας FTA με την Ταϊλάνδη, ας πούμε τη Μαλαισία και κάνει κανείς εισαγωγή από την Ταϊλάνδη τη Μαλαισία, κατά πόσο δηλώνεται στην εξαγωγή στην Ευρώπη το κράτος ως προερχόμενο από τη Μαλαισία ή από την Ταϊλάνδη είναι σημαντικό στατιστικά. Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το ποστό του εμπορίου μας με την Μαλαισία ή την Ταϊλάνδη. Αλλά δεν επηρεάζει αυτό την αντιμετώπιση του αυτοκινήτου εντός της Ένωσης. Ε, αφού έχουμε τους δασμούς του πλέον ευνοούμενου κράτους. Αυτό είναι μια απλή εικόνα της κατάστασης για τις ορισμένες περιπτώσεις. Μπορούμε να εφαρμόσουμε άλλα μέτρα ε, αντι για παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο μέλος του ΠΟΕ και εκεί το ζήτημα της καταγωγής ε, έχει μεγαλύτερη σημασία και εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις ε, μη προτιμησιακός κανένας καταγωγής στον ΠΟΕ γίνονται προσπάθειες για να επιτευχθεί μια συμφωνία για τους μη προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής για διάφορους τύπους προϊόντων. Οι εργασίες αυτές τρέχουν εδώ και 21 χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Ε, το χρονικό διάστημα αυτό εξηγείται από την πολυπλοκότητα της άσκησης. Ε, μετά έχουμε το προτιμησιακό εμπόριο με προϊόντα διαφόρων χωρών να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Αν το προϊόν προέρχεται από το Βιετνάμ όπου έχουμε FTA ή αν έρχεται από τη Μαλαισία με την οποία δεν έχουμε, εκεί κάνουμε τη διαφορά. Και αυτό επηρεάζει τον τρόπο αντιμετώπισης του προϊόντος κατά την εισαγωγή του. Οι προτιμησιακοί κανόνες εισαγωγής, ε, α, ε, καταγωγής αποτελούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Λόγω της ε, ε προτίμησής μας προς την ανάπτυξη γενικότερα, που είναι προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη, θέλουμε να ξέρουμε ένα προϊόν στο οποίο έχουμε χορηγήσει προτιμησιακή αντιμετώπιση, κατά πόσο πράγματι Θέλουμε να ξέρουμε αν είναι ένα προϊόν ε, το, το, και υπό ποιες συνθήκες παράγεται. Και μετά έχουμε όλο και περισσότερες συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών όπου, υπάρχει προτιμησία, όπου εφαρμόζονται προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής. Ο αριθμός τους αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον. Οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής ε, γίνονται όλο και πιο σημαντικοί στο σύστημά μας. Και όπως είπε και ο συναδέλφος ε, κ. Σάλμπερ, σταδιακά εξορθολογίζουμε την προτιμησιακή διευθέτηση που έχουμε. Το 2011 είχαμε τον νέο κανονισμό ε, ESP, όπου απλουστεύσαμε τους κανόνες κατά προϊόν, τους κανόνες που έχουμε για κάθε προϊόν για να ορίζουμε από πού προέρχονται. Επίσης απλουστεύσαμε τον τύπο εξαγωγέων που μπορούν να υποφεληθούν από την προτίμηση και χρησιμοποιήσαμε και κάποιες διαδικαστικές απλουστεύσεις εκεί. Όλα αυτά αποτυπώνονται στις ε, επερχόμενες ε, ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών που είχαμε. Εφαρμόζουμε τους ίδιους κανόνες προτιμησιακούς για όλες τις συμφωνίες. Όχι. Οι προτιμησιακοί κανόνες ε, Συνήθω αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων και είναι και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της δικής μας προσέγγισης. Όπως βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, του πιο χαλαρούς κανόνες καταγωγής τις έχουμε με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, επειδή θέλουμε να ευνοήσουμε τις εξαγωγές από αυτές τις χώρες προς την Ένωση για, με σκοπούς αναπτυξιακούς και μετά, σας ξαναλέω, όλα αυτά είναι απλουστευμένα. Ε, διότι η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Αλλά γενικά το 70% των μη ε, προερχόμενων ε, υλικών τα επιτρέπουμε. Μόνο το 30% της αξίας είναι εγχώρια. Για τους δικαιούχους των γενικευμένων συστήματος προϊόντων επιτρέπουμε το πολύ 50% υλικών που δεν προέρχονται από τη χώρα. Με τις FTA επίσης εκεί προσπαθούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ των FTA με αναπτυγμένες χώρες όπου επιτρέπουμε ανάπτυξη του προϊόντας με 50 ως 60% προϊόντων που δεν είναι της χώρας ε, και μετά έχουμε τις FTA με ανεπτυγμένες χώρες ε, όπου το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό αυτό, αυτό είναι 45 με 50% το ποσοστό αυτό των μη καταγόμενων υλών. Ε, οπότε όλα αυτά εξαρτώνται όχι μόνο από την βούλησή μας ε, ε χρειάζονται πάντα διαπραγματεύσεις ε, ε, και ακόμη και αν έχουμε μια γενική προσέγγιση με μια χώρα, τι διαπραγματευόμαστε κατά προϊόν με τους εταίρους μας. Γενικά φέρνει αποτελέσματα. Πρόσφατα εκδόθηκε μια έκθεση που συγκρίνει τις τις και καθεστώτα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσματα είναι καλά. Έχουμε την ε, μεγαλύτερη χρήση των προτιμήσεων και έχουμε ε, καλό σύνολο προτιμήσεων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών λειτουργεί. Για τις ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση. Κατά μέσο όρο χρησιμοποιούνται οι προτιμήσεις κατά 80% αυτές που έχουν χορηγήσει σε τρίτες χώρες. όλα εξαρτώνται και από τους τομείς την, ε, όπως εξειδικευμένες είναι οι εξαγωγές του κάθε κράτους κράτους. Now, do we with rules of to, uh, Συμβάλλουμε με τους κανόνες καταγωγής ε, στην ανάπτυξη παγκοσμίω. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε και να μην δημιουργούμε πρόβλημα. Ένας λόγος για τον οποίο χαλαρώσαμε τους κανόνες καταγωγής μετά από τη μεταρρύθμιση των GSP στις FTA μας. Αυτό προσπαθεί να αποτυπώσει στις FTA μέχρι τώρα. Έχουμε μέχρι το πολύ 50 έως 70% ξένα υλικά σε ένα προϊόν ώστε να υπόκειται στην FTA. Ενώ στην προ... Ε, στις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών πρώτης γενιάς με τη Χιλή ή το Μεξικό για παράδειγμα είχαμε πιο περιοριστικά όρια 30-40% μη καταγόμενων υλών. Ήμασταν πολύ περιοριστικοί κατά την αναθεώρηση στη διαπραγμάτευση που έχουμε τώρα με το Μεξικό. Θα επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα, θα τα εξετάσουμε κατά πώ θα χαλαρώσουμε του κανόνε καταγωγή για διάφορα προϊόντα, ώστε να αποτυπώνεται το γεγονό ότι οι φορεί μα τώρα ε, είναι πιο ολοκληρωμένοι και χρειάζονται περισσότερα ε, ξένα υλικά για να παραγούν. Ε, κάτι που συμβαίνει και στους δικούς μας παραγωγούς και στους εταίρων μας. Όταν έχουμε μια συμφωνία με την Κορέα, για να είναι ένα αυτοκίνητο ευρωπαϊκό υπολογίζουμε τα εξαρτήματα που προερχόνται από την Κορέα και συναρμολογούνται στην Ευρώπη σαν ευρωπαϊκό ε, αυτοκίνητο όσο και τα ευρωπαϊκά εξαρτήματα ώστε να καθορίσουμε κατά πόσο είναι ευρωπαϊκό ένα αυτοκίνητο έχουμε αυτή τη σώρευση δηλαδή με τους εταίρους και έχουμε και περιφερειακή σώρευση ειδικότερα με τους κανόνες καταγωγής ε, πανευρωμεσαγειακής ε, σόρευσης. Ο, προσπαθούμε να έχουμε τη σόρευση με τους, γειτόνες, με τους γειτονές μας. Αυτό είναι ε, κρίσιμο για ορισμένους τομείς όπου όταν έχουμε ας πούμε στην κλωστοβιφαντουργία παράγεται το ύφασμα στην Ευρώπη ενώ η επεξεργασία γίνεται από μια εταίρο χώρα και μετά το προϊόν έχει καταγωγή περιφερειακή. Και έτσι συμβάλλουμε στην ενίσχυση των παγκόσμιων ε, αλυσίδων αξίας, ειδικότερα στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας. Επίσης προσπαθούμε να απλουστεύσουμε, όπως είπε ο συνάδελφός μου, να απλουστεύσουμε τη διαδικασία με μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων ε, συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών. Προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, απομακρυνόμαστε από τα επίσημα πιστο, τελωνιακά πιστοποιητικά σε πιστοποιητικά πώληση των εξαγωγέων, απομακρυνόμαστε από τους εγκεκριμένους εξαγωγείς, κάτι που ήταν πολύ πιο περίπλοκο για τους εξαγωγείς το να εγγραφούν ως εγγεγραμμένοι εξαγωγείς ε, στη σχετική βάση δεδομένων, όπου ένας εξαγωγέας μπορούσε να έχει ευκολότερη πρόσβαση ε, Απολαμβάνοντα έτσι πιο εύκολα ε, το προτιμησιακό καθεστώς μιας FTA. Συμπερασματικά έχουμε μια κατάσταση όπου εμείς ε, χρειάζεται αφενός να εστιαστούμε στους προμηθησιακούς κανόνες. Οι μη προτιμησιακοί δεν μας απασχολούν αυτή τη στιγμή τόσο πολύ. Οι προτιμησιακοί κανόνες ε, απαιτούν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του να καθορίσουμε την καταγωγή στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένη συμφωνίας ελευθερών συναλλαγών ή στο πλαίσιο ενό συστήματος ωφελών ε, και μεταξύ της πολυπλοκότητας των διοικητικών απαιτήσεων. Ε, επίση, προσπαθούμε να επιτύχουμε και κάποια χαλάρωση. Εξαρτάται από του εταίρου και τα προϊόντα. Λαμβάνουμε υπόψη επίση και πιθανές αλλαγές, επιτρέποντας σόρευση ε, σε διμερή βάση και προσπαθούμε να προστέύσουμε τις διαδικασίες για την πρόσβαση στο προτιμησιακό καθεστώς. Ε, φυσικά τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε πολλές πληροφορίες ε, σχετικά με αυτό το πολύπλοκο σύστημα. Έχετε τώρα τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις. Μαρία Αρένα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ περίπλοκο ζήτημα, πράγματι, και φαίνεται πολύ τεχνικό. Συγχρόνω, όμως εγώ πιστεύω ότι είναι και αρκετά πολιτικό. Και αυτά τα τελευταία που μας είπατε, αυτό ακριβώς δείχνουν. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι μια στρατηγική που ζητάει ζητάει να ε, δέχεται η Ευρώπη προϊόντα που όλο και περισσότερο ε, παράγονται αλλού ή που όλο και περισσότερο παράγονται στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολιτικό το ζήτημα όσον αφορά τη στρατηγική μας. Έχω διάφορες ερωτήσεις που είναι, για παράδειγμα, είπατε ότι πρέπει να τροποποιηθεί το σύστημα για να είναι πιο αποτελεσματικό, αλλά να κρατήσουμε τον στόχο του κανόνα καταγωγής. Υπάρχει και το θέμα των ετικετών και το θέμα της πράλευσης ενός προϊόντος, γιατί εσείς ασχολείστε και με την ετικέτα όταν ασχολείστε με τον κανόνα καταγωγής. Πώς λοιπόν αυτά τα δύο τα συνδυάζουμε μαζί. Δεύτερον, Μιλήσατε για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πράγματι, στις συμφωνίες που έχουμε με την Αφρική υπάρχει κάποια ευελιξία όσον αφορά τον κανόνα καταγωγής για την ε, πτυχή της συσσόρευσης, δηλαδή από διάφορες αφρικανικές χώρες και όχι από μία μόνο. Πώς να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να συμμορφωθούν με τον κανόνα καταγωγής. Ξέρετε ότι λίγες χώρες εκεί μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες, πώς να τους βοηθήσουμε διοικητικά, ε, στα τελωνία για να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Τρίτον, δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα της μη προτίμησης. Μιλήσαμε για την προτίμηση για τα πλέον ευνούμενα κράτη, όχι για τα μη ευνούμενα κράτη. Στα κατεχόμενα, για παράδειγμα, πώς διαχειρίζεστε αυτό το θέμα για τον κανόνα καταγωγής. Το θέμα των ετικετών έχει τεθεί. Πού βρισκόμαστε λοιπόν και στην ε, Δυτική Σαχάρα πάλι υπάρχει ζήτημα γιατί έχουμε αυτή τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Μαρόκο. Άρα το θέμα της καταγωγής έχει να κάνει με προϊόντα τα οποία παράγονται σε δάφη τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα κανονικά από την Ευρώπη. Τι κάνετε για αυτές τις περιπτώσεις. Και έχω και πολλά ερωτήματα όσον αφορά την αυτοπιστοποίηση. Και αυτό έχει να κάνει με τα καταχώμενα εδάφη. Το Ισραήλ αυτοπιστοποιεί την καταγωγή. Αλλά υπάρχει πρόβλημα όμως γιατί υπάρχουν προϊόντα τα οποία ε, παράγονται στη Δυτική Όχθη. Οπότε τίθεται υπομφισβήτηση το καθεστώς αυτό της αυτοπιστοποίησης σε αυτή την περίπτωση. Και τι κάνουμε, σταματάμε τη διαδικασία μέχρι να γίνει ο έλεγχος. Εσείς είπατε ότι όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία είναι η χώρα που εισάγει που πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση. Ναι, αλλά προβλέπονται διαδικασίες παύσης, αναστολής, γιατί αν η εξολόγηση κρατήσει 10 χρόνια θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την προτιμησιακή κατάσταση περιμένοντας τα αποτελέσματα. Οπότε δίνουμε στους ανταγωνιστές το κλειδί για να αυτοπιστοποιούνται. Χωρίς να διαθέτουμε εμείς τα μέσα να προχωρήσουμε σε αναστολή του καθεστώτος αυτού όσο γίνεται μια αξιολόγηση. Και εντάξει, φαντάζομαι έχουν και άλλοι ερωτήσει οπότε θα σταματήσω εδώ. Ακριβώ. David. Ευχαριστώ. Σε κάποιο βαθμό η Μαρία αναφέρθηκε σε ένα θέμα που ήθελα να θίξω και εγώ, την αυτοπιστοποίηση. Έχει νόημα να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, αλλά υπάρχει και αρκετή απάτη. Και αναρωτιέμαι, εάν η χώρα εισαγωγή διαπιστώσει, η ευρωπαϊκή χώρα εισαγωγή έχει διαπιστώσει ότι ε, έχει λάθος επισήμανση το προϊόν. Μπορούμε να εφαρμόσουμε τελωνιακές διαδικασίες, μπορούμε να κάνουμε κάτι μέχρι να διαπιστώσουμε εάν είναι σωστή η επισήμανση ή υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Ήταν χρήσιμη η διαφάνεια διότι δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στα διάφορα προτιμησιακά καθεστώτα, αλλά... Μήπως υπάρχει αντικίνητρο ε, στο να μεταφερθεί κανείς ε, από το ένα καθεστώς στο άλλο, προς ένα καθεστώς δηλαδή ελεύθερο εμπορίου. Αυτό πιθανότητα, πιθανότατα να είναι πιο περιοριστικό από ότι οι κανόνες ε, καταγωγής. Και επίσης, όσον αφορά την περιφερειακή συσσόρευση, είναι αυτό πιο δυνατό να γίνει με μια ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου από ότι με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και τι γίνεται με τις χώρες που εμπίπτουν στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων αλλά έχουν γειτονικέ χώρες που δεν εμπίπτουν στο καθεστώς αυτό. Έτσι μπορεί κάποιες χώρες να βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Πώς ε, αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Και τέλος, όσον αφορά τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, αν δεν κάνω λάθος, και σε σχέση με το Βιετνάμ είπαμε ότι ε, προϊόντα κλωστοφαντουργίας από την Κίνα δεν μπορούν να, να συμπεριληφθούν. Ε, με, για την Ινδονησία τι ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σάινφελτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, δύο ερωτήσεις έχω. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε εδώ δύο διαφορετικά επίπεδα. Έχουμε το νομικό επίπεδο και το ε, πραγματικό επίπεδο. Τι εννοώ όταν λέω νομικό επίπεδο. Τους κανόνες ε, που καθορίζουν την καταγωγή. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι και προβλέπονται διαφορετικά προτιμησιακά καθεστώτα. Θα πρέπει φυσικά να λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό οι κανόνες καταγωγής. Αλλιώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν υπάρχει προτίμηση λόγω της καταγωγής ή όχι. αν ξεφύγουμε από το νομικό επίπεδο, τίθεται το ερώτημα στο πλαίσιο του παγκοσμίου εμπορίου. Σε όλο τον κόσμο γίνονται επενδύσεις, παράγονται προϊόντα. Το προϊόν ε, αποτελείται από ε, τμήματα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές υπήρους μερικές φορές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν τίθεται το ερώτημα εάν έχουν νόημα οι κανόνες καταγωγής. Θα με ενδιαφέρε η απάντηση στο ερώτημα αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια στρατηγική για το μέλλον. Και μια δευτερεύουσα ερώτηση όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ συχνά ένα προϊόν, λέω για παράδειγμα τώρα, προέρχεται από την Τσεχία, περιέχει όμως τμήματα από τη Γερμανία, τη Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο και τίθεται το ερώτημα αν το προϊόν αυτό είναι γερμανικό, βρετανικό ή τσεχικό. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα πρέπει να λέει κανεί ότι είναι ε, προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όχι συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ε, υπάρχει και μία νομική και οικονομική διαμάχη πάνω στο θέμα αυτό και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη θέση σας. Τελευταία παρατήρηση. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Μίλησα για το νομικό επίπεδο, αλλά τώρα φτάνουμε στο πραγματικό επίπεδο. Ένας πολίτης λοιπόν αγοράζει ένα προϊόν. Ο πρόεδρος μας είναι Γερμανός, οπότε θα χρησιμοποιήσω γερμανικό παράδειγμα. Ένας Γάλλος αγοράζει στη Βαβαρία, στη Γερμανία δηλαδή, την αγοράσει εκεί. Ε, μια BMW. κατασκευασμένη στις Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα λοιπόν τι έχει αγοράσει, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, γερμανικό ή ε, αμερικάνικο. Ο Χέλμουτ Σόλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους ομιλητές μας για την εισαγωγή σε αυτό το πολύπλοκο θέμα και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είχα τις ίδιες ερωτήσεις με τον ε, συνάδελφο ε, Σάινφελτ. Μιλήσατε για την ε, εθνικότητα ενός προϊόντος και στην παγκόσμια οικονομία τίθεται το θέμα αυτό. Παράδειγμα, ένα smartphone που περιέχει κομμάτια που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χώρες. Πώς καθορίζεται λοιπόν ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Ιαπωνία. Ο καταναλωτής πώς μπορεί να το γνωρίζει αυτό και πώς καθορίζουμε την καταγωγή του προϊόντος στη στιγμή που αποτελείται από τμήματα κατασκευασμένα σε διάφορες χώρες. Αυτό συνδέεται και με αυτά που καθορίζουμε στις διμερείς μας εμπορικές συμφωνίες. Στον τομέα της γεωργίας ε, συμφωνούμε πάνω σε ισχυρμένε ποσότητες. Ε, τι ισχύει για παράδειγμα για τις μπανάνες. Έχουμε διάφορες αλυσίδες μέσω των οποίων προμηθεύονται αυτές οι μπανάνες. Οι κανόνες καταγωγής πώς επηρεάζουν την προσφορά των προϊόντων για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιθανότατα να συνδέεται και με το θέμα της αυτοπιστοποίησης, ε, σίγουρα συνδέεται με το θέμα της επισήμανσης. Τελικά όμως, στις διαπραγματεύσεις, η διαμάχη έχει να κάνει με το αν τελικά θα επιλέξω 60 τόνους μπανάνες τσικίτα ή ε, μπανάνες από χώρες ΑΚΕ. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τους κανόνες καταγωγής, πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε, διαφων... σε διαφανείς διαδικασίες ε, οργάνωσης της αγοράς μας. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, δύο ερωτήσεις από μένα. Καταρχάς, Αχέκη μου ανέφερε σχετικά με τα διαφορετικά επίπεδα και τα διάφορα όρια ε, των κανόνων καταγωγής. Ε, όλα αυτά μοιάζουν με μια μακαρονάδα. Ε, και αν αναφερθώ στο λιμάνι που γνωρίζω καλύτερα, το λιμάνι του Αμβούργου, όπου καταφθάνουν πολλά κοντέινερ, πώς μπορούν οι τελωνιακοί αξιωματούχοι να ελέγξουν αυτή, να εξετάσουν αυτή τη μακαρονάδα με βάση την πραγματικότητα, τα πραγματικά προϊόντα ή με βάση έγγραφα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να μπορεί να γίνει σωστός έλεγχος του συστήματος αυτού. Και δεύτερον, ο κύριος Σάινφελντ ανέφερε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει απόφαση σχετικά με τους κανόνες καταγωγής. Στη Βρετανία τι θα γίνει. στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μόνο το 40% για παράδειγμα μπορεί να προέρχεται από τη το Ηνωμένο Βασίλειο, το υπόλοιπο από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τους κανόνες αυτούς. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω και να συμπληρώσω και κάποιες πληροφορίες για την επισήμανση. Την καταγωγή πρέπει να τη γνωρίζει κανείς σε μια προτιμησιακή συμφωνία. Όταν μπει πέρα στα σύνορα χρειαζόμαστε μια διασάφηση που να αναφέρει την καταγωγή του προϊόντος στο τελωνίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν απαιτεί ετικέτα η επισήμανση. Αυτό είναι που, σημαντικό, που είναι σημαντικό είναι η διασάφηση εισαγωγή να είναι σωστή ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές ποια είναι η καταγωγή του προϊόντος του συνόλου του και των συστατικών του, των εξαρτημάτων του. Όπως είπε ο κ. Σόλτς, το ανοίγει κανείς και βρίσκει διάφορα εξαρτήματα, για παράδειγμα σε ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά μπορεί να έχουν μια ετικέτα καταγωγής και άλλα όχι. Αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο πράγματα, την επισήμανση και ποια καταγωγή θεωρείται ότι έχει κατά την εισαγωγή ένα προϊόν. Στι συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών μα συνήθω ε, ζητάμε από του εταίρου μα, ε, αν αυτοί απαιτούν ε, επισήμανση τη καταγωγή επειδή δεν το απαιτούν όλες οι χώρες. Αν εσεί λοιπόν στη χώρα σας τους λέμε απαιτείτε επισήμανση των προϊόντων στην επικράτειά σας παρακαλούμε επιτρέψτε πέραν της ετικέτας ε, Made in France, Made in ε, Germany να υπάρχει η ετικέτα Made in the EU. Αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό σημείο για μας όταν είναι υποχρεωτική επισήμανση για προϊόντα στην χώρα εταίρο μας. Πώς βοηθάμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, για τα θέματα καταγωγής. Έχουμε ένα σχετικά χαλαρό κανόνα. 70% μη καταγόμενα υλικά για τις ε, ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες είναι χαλαρός κανόνας. Μετά έχουμε τον κανόνα της όρευσης. Στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρική σχέσης επιτρέπουμε τη σόρευση και μεταξύ των συμφωνιών εταιρική σχέσης, δηλαδή με εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για παράδειγμα, γίνεται μια προσπάθεια να επιτρέπεται η σώρευση μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών ε, με EPA για τους κανόνες καταγωγής. Επίσης προσπαθούμε να αναπλουστεύσουμε τις διαδικασίες από την έγκριση των εξαγωγέων της άλλης πλευράς έχουμε περάσει στο μητρό των εξαγωγέων που είναι λιγότερο γραφειοκρατικό. Προσπαθούμε λοιπόν να απλουστεύσουμε τα διαδικαστικά και να χαλαρώσουμε τους κανόνες, καθώς και να ενισχύσουμε την, τις δυνατότητες σώρευσης. Μετατίθεται το ζήτημα του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και των ε, συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών. Χάνει κανείς ή κερδίζει. Είσαι το Βιετνάμ. Θες να μείνεις εκεί που ήσουν ή θες να περάσεις σε μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών. Το Βιετνάμ το έπραξε. Υπάρχουν πλέον εκτήματα. Πρώτα απ' όλα η FTA είναι μία μόνιμη συμφωνία επί της αρχής. Μπορεί να υπόκειται σε έναν μηχανισμό αναθεώρησης, αλλά είναι διμερής αυτός. Ενώ η... το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι μια μονομερής ε, ε, παραχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ε, αν μια μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πιο αυστηρούς κανόνες της, ή αν αναπτυχθεί η αν χωρα σου μπορεί να μην εντάσσε πλέον στο, στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων γιατί δεν θα πληρούνται πλέον οι κανόνες ενώ στην FTA υπάρχουν, είναι διμερές η συμφωνία Κάποια στοιχεία σώρευσης τώρα, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Βιετνάμ είχαμε μια σώρευση, δεν είχαμε μια σώρευση, συγγνώμη, αλλά, γενική, αλλά είχαμε μια σώρευση ε, για τα ε, υφάσματα με την Κορέα ναι, επειδή αυτό τους ενδιαφέρε. Γιατί η φαντουργία τους ε, ε, έχει σχέση με τη γενική φαντουργία. Οπότε έχεις κάποιο συμφέρον ε, να περάσει κανείς από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων στην FTA. Ας δούμε την περίπτωση της Σιγκαπούρης όπου διατηρούμε την περιφερειακή σώρευση με τις χώρες ΕΣΕΑΝ. κλωστοϊφαντουργία στην Κίνα δεν κατάλαβα καλά. Για την περίπτωση του Βιετνάμ επιτρέπουμε σόρευση ε, ε, στα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα με την Κορέα. Αλλά δεν επιτρέπουμε τη σόρευση με την, με την Κίνα. Η διαδικασία αποδοχή τη όρευση σε μια FTA μα επιτρέπει να στοχεύσουμε και το τι κάνουμε όσον αφορά τη χαλάρωση των κανόνων. Όταν προσπαθούμε να χαλαρώσουμε του κανόνε ε, για παράδειγμα περνώντας από 50% ξένων μη καταγωμένων υλικών σε 70% αυτή η διαφορά του 20% επιτρέπεται να συμπληρωθεί από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ενώ αν παραμείνουμε στο κατόφλι του 50% των μη καταγωμένων υλών και επιτρέπουμε σώρευση με μία χώρα ή μια άλλη, ε, εκεί στοχεύουμε κάπως περισσότερο το άνοιγμα που επιτρέπουμε στο προϊόν τους. Στην περίπτωση των κλωστοφαντουργικών το Βιετνάμ ε, είχε στοχευθεί μόνο όσον αφορά την Κορέα. Συγγνώμη, η ερώτησή μου ήταν θα έχουμε την ίδια ρήτρα για την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά. Βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη διαδικασία. Δεν έχουμε υποβάλει ακόμα κείμενο για την Ινδονησία ή τις Φιλιππίνες. και εκεί θα τεθεί αυτό το ζήτημα που μπορεί να συζητηθεί ή όχι στις διαπραγματεύσεις ε, βάσει αιτήματος Ινδονησίας ή Φιλίππινων. Για το ζήτημα των κανόνων καταγωγής έχουν νόημα. Ναι, έχουν νόημα ε, στην περίπτωση προτιμησιακών συμφωνιών. Αν τα ταραβήξουμε τα πράγματα στα άκρα και έχουμε μια FTA με μια χώρα χωρίς κανένα κανόνα καταγωγής για... Η συμφωνία αυτή ελευθέρωση συναλλαγών θα είναι απλά μονομερής ε, απελευθέρωση με όλες τις χώρες του κόσμου, διότι οτιδήποτε παράγεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα μπορούσε να διοχετευτεί μέσα αυτής της χώρας. Αν έχουμε λοιπόν μια συμφωνία με την χώρα Χ, χωρίς κανόνες καταγωγής, ουσιαστικά οτιδήποτε μπαίνει από αυτή τη χώρα θα υπόκειται στο προτιμησιακό καθεστώς, οπότε ε, έτσι θα μπορούσε να πολύ μια χώρα όλες τις εξαγωγές της. αν, πάρουμε μια, αν λάβουμε μια άλλη ακραία θέση και πούμε ότι μονομερός απελευθερώνουμε όλο μας το εμπόριο και μηδενίζουμε όλους τους δασμούς, σε αυτή την περίπτωση θα χρειάζονταν FTA στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Union. Do we care if the is uh, Στην Ένωση μας ενδιαφέρει αν ένα προϊόν είναι τσεχικό ή γαλλικό. Είναι θέμα αντιμετώπισης και επισήμανσης. Η επισήμανση είναι ένα ζήτημα που αντιμετώπιση και καιρό χωρίς πρόοδο. Η ζήτηση της αντιμετώπισης όμως ε, και της επεξεργασίας δεν έχει σημασία το σημαντικό είναι να έχουμε τον έλεγχο στα σύνορα και να εφαρμόζουμε του δασμού στα σύνορα. Εφόσον μπει σε ελεύθερη κυκλοφορία ένα υλικό, ένα προϊόν στην Ένωση, είτε έχει συναρμολογηθεί, το να συναρμολογηθεί στη Γαλλία ή στην Τσεχία δεν έχει σημασία. Θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο στην Ένωση. Οπότε το ερώτημα για εμά είναι κατά πόσο έχουμε ένα γερμανικό ή ένα αμερικανικό αυτοκίνητο. Το ζήτημα το, το αυτοκίνητο είναι γερμανικό-αμερικανικό ε, ε τίθεται όταν μπαίνει ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, για να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστεί δασμός. Ε, τώρα, το τι κάνουμε λογικά ή συναισθηματικά, αν προτιμάμε ένα προϊόν που έχει παραχθεί στη χώρα μας ή κάπου αλλού, Εκεί είναι το θέμα. Αλλιώ, ε, εφόσον έχει μπει στην Ένωση, δεν έχει διαφορά. Κάποιο προϊόν μπορεί να κινηθεί παντού. Τα έξυπνα τηλέφωνα είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα. Υπόκειται σε μια άλλη συμφωνία, δεν εφαρμόζουμε δασμού για τα smartphone. Αν έπρεπε για ένα προϊόν που υπόκειται σε κανόνε καταγωγή, τότε ε, η καταγωγή και η επισήμανση δεν χρειάζεται να συνδέονται. Για τι μπανάνες, κανονικές μπανάνες ξέρουμε την καταγωγή, δεν έχει συστατικά, δεν έχει εξαρτήματα, κάπου παράγεται η μπανάνα, ε, υπάρχουν κάποια λιπάσματα και τα λοιπά φυτοφάρμακα, αλλά αυτά είναι τα υλικά που χρησιμοποιείται στην παραγωγή της μπανάνας. Ε, ξέρουμε που είναι τα δέντρα όμως και ξέρουμε που ε, έχει παραχθεί μια μπανάνα. Πρέπει να ότι την παρανόηση από τα Κανάρια νησιά φυσικά είναι πιο γευστικές, αλλά υπάρχουν ε, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο ε, και ο έλεγχος είναι διαφορετικός. Θα το εξηγήσουμε πιο λεπτομέρως αργότερα. The control is not... Ο έλεγχος έχει να κάνει με το σύνολο, με την αρχή της προτιμησιακής μεταχείρισης αλλά έχει να κάνει και με το θέμα της ασφάλειας. Οι έλεγχοι στα σύνορα γίνονται βάσει αξιολόγησης κινδύνου, πληροφοριών κτλ. Ο όγκος του εμπορίου που έρχεται από τον Βούργο ή από το Ρότερνταμ είναι τόσο μεγάλος που δεν είναι δυνατόν να ανοιχτεί κάθε κοντέινερ και να ελεγχθεί. Στατιστικά υπάρχει ένα επίπεδο, ο Άλβερ θα τα πει καλύτερα, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο ελέγχεται. Μικρό ποσοστό, γιατί είναι τεράστιος όγκος του εμπορίου. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, όπως είναι ο κίνδυνος. Επιτρέψτε μου τώρα να μην απαντήσω για το θέμα του Brexit. Πάντως οι κανόνες που διαθέτουμε και τόπο όταν σας έδειξα τη διαφάνεια με τα διάφορα ποσοστά που εφαρμόζουμε για διαφορετικού είδους ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή γενικευμένων προτιμήσεων. Εξαρτάται λοιπόν από το προϊόν, από τις διαπραγματεύσεις και υπάρχουν και ειδικοί κανόνες προϊόντος που μας οδηγεί στο ένα ή στο άλλο ποσοστό. Όπως επίσης είπα, όταν έχουμε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ε, Κορέα, για παράδειγμα, έχουμε και συσσόρευση προέλευση. Σε διαφορετικό βέβαια επίπεδο, αλλά πρέπει να το απλοποιήσουμε. Αν έχουμε μια συμφωνία με την Κορέα και η Κορέα συναρμολογεί ένα αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιεί εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυτά τα εξαρτήματα που εξήχθησαν από την Ευρώπη στην Κορέα είναι μέρος του ποσοστού των υλικών καταγωγής. Και ανάλογα μπορεί και η Κορέα να αποκτήσει λοιπόν το καθεστώς αυτό καταγωγής ή όχι για το συγκεκριμένο προϊόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ σε δύο πτυχές μόνο η μία έχει να κάνει με τον έλεγχο, όπως είπατε, και η άλλη έχει να κάνει με τα δάφη της Δυτικής Σαχάρας και της Δυτικής Όχθης. Και θα έρθω και σε κάποια στοιχεία που αναφέρθηκαν όπως οι ετικέτες και η αυτοπιστοποίηση. Έρχομαι πίσω στην διάκριση των κανόνων του πλέον ευνοούμενου και του μη πλέον ευνοούμενου εταίρου. Βασιζόμαστε σε κανόνες, όπως ε, σας είπα, που έχουν να κάνουν ε, με την χώρα εισαγωγέα. Εδώ δεν πρόκειται για διεθνείς προδιαγραφές. Αποφασίζει αυτός που εισάγει. Δεύτερον, το θέμα της ε, αυτοπιστοποίησης δεν παίζει στο θέμα των μη πλέον ευνοούμενων εταίρων. Τότε η απόδειξη της προέλευσης του προϊόντος καθορίζεται από τον εισαγωγέα. Το πώς αποδεικνύεται δηλαδή η προέλευση ενός προϊόντος. Δεν έχει να κάνει με μια συμφωνία. Όταν όμως μιλάμε για την Δυτική Σαχάρα και για την Δυτική Όχθη, εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερα με το θέμα της προτιμησιακής μεταχείρισης στις συμφωνίες που έχουμε με το Μαρόκο στην περίπτωση και με το Ισραήλ στην άλλη. Και βέβαια το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα εδάφια αυτά. Πώς τα θεωρούμε. Τι θεωρούμε ότι είναι επικράτεια του Μαρόκου και του Ισραήλ. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που τίθεται. Μπορούμε να εφαρμόσουμε προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα τα οποία παράγονται στη Δυτική Όχθη. Η απάντηση είναι όχι. Μπορούμε να έχουμε προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Και πάλι η απάντηση είναι όχι. Γιατί σύμφωνα με το δικαστήριο, τα εδάφια αυτά δεν καλύπτονται από τις συμφωνίες που έχουμε με τις χώρες αυτές, Μαροκό και Ισραήλ. Είναι το μόνο που μπορώ να πω. Όσον αφορά τώρα τους ελέγχου, τα είπε και ο λίγο, όταν τα τελωνία ελέγχουν την ε, προέλευση, την προτιμησιακή ενός προϊόντος, έχουμε διάφορα εργαλεία. Το ένα είναι η αυτοπιστοποίηση, έτσι, το πιστοποιητικό που εκδίδει η ίδια η χώρα που εξάγει και που βεβαιώνει την καταγωγή του προϊόντος. Αλλά υπάρχουν και επιπλέον πληροφορίες από ε, μυστικές πληροφορίες που έχουμε από έρευνες, αναλύσεις που κάνουμε όσον αφορά την προέλευση του προϊόντος. Και εδώ πάμε πίσω στο σύστημα του ελέγχου. Δηλαδή πώς εφαρμόζονται οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Πάμε πίσω στο σύστημα επαλήθευσης. Σας είπα πριν για την επαλήθευση μέσω διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των μερών υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης. Έχουμε συμφωνίες και οι σχετικές διατάξεις έχουν συμπεριληφθεί πολλές φορές στις συμφωνίες ελεύθερου μπορείου. Και τέλος υπάρχουν και κυρώσεις. Αν ισχυριστείς κάτι το οποίο δεν ισχύει, τότε υπάρχει δυνατότητα, μάλλον να το πω αλλιώς, αν πιστοποιήσεις με έναν τρόπο το προϊόν σου, περιμένεις και κυρώσεις αν τελικά η δήλωση αυτή δεν είναι ορθή. Και αν ε, ισχυριστεί κάτι το οποίο δεν ισχύει, επίσης υπάρχει δυνατότητα κυρώσεων. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δυνατότητες που έχουμε για να έχουμε ένα αποδεκτό επίπεδο συνέπειας από πλευράς των χωρών που εξάγουν. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας. Θα είμαστε σε επαφή σχετικά με το θέμα αυτό, διότι το θέμα της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και τη συμπερίληψη των κανόνων αυτών σε μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίε μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, και αναφέρομαι και ε, σε ενδεχόμενη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά που ακούσαμε ήταν λίγο πολύ η εικόνα εκ των έσω. Τώρα θα καλέσουμε εξωτερικούς προσκεκλημένους που θα μας μιλήσουν για τους κανόνες καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν δύο εμπειρογνώμονες, τον Τόμας Βλωστόφσκι και την Άννα Γερζεύσκα. Ο Τόμας Βλωστόφσκι ε, έρχεται από την Trade Defense, ενώ η Άννα Γερζεύσκα είναι εμπειρογνώμων πάνω στις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Θα ήθελα λοιπόν να τους καλέσω να μας δώσουν την εξωτερική, μια εξωτερική άποψη ε, πάνω στον κανονισμό μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Τόμας Βλωστόφσκι, είμαι νομικός, ασχολούμαι με την πολιτική εμπορίου εδώ και 14 χρόνια, εργάζομαι στις Ηνωμένε Πολιτείε και τα νέα τελευταία χρόνια εργάζομαι εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις αναλυτικές ε, σκέψεις μου πάνω στους κανόνες καταγωγής. Ε, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τέσσερα θέματα. Ε, ένα στο οποίο μάλλον δεν χρειάζεται να επικεντρωθούμε πάρα πολύ είναι το πώς οι κανόνες καταγωγής είναι σημαντικοί. Διότι οι κανόνες καταγωγής είναι η μηχανή στο εμπόριο. Ε, και τα πλεονεκτήματα των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα μείωση των δασμών. Αν δεν καταλάβουμε όμω πώ λειτουργούν οι ε, κανόνε καταγωγή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι ε, συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα τα οποία είναι χρήσιμο να σκεφτείτε κατά την εξέταση των κανόνων καταγωγής. Ποιος επωφελείται και τέτοιες συζητήσεις θα πρέπει να κάνετε, διότι αυτή τη στιγμή αυτά τα θέματα βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά ε, στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τρίτο θέμα συνδέεται με το δεύτερο, η διαδικασία, οι κανόνες καταγωγής αυτοί από που προέρχονται και πώς μπορούμε να τους επηρεάσουμε, να τους τροποποιήσουμε και ε, τέταρτον, αν έχω λίγο χρόνο παραπάνω, θα ήθελα να μιλήσω για το πιο συναρπαστικό θέμα αυτή τη στιγμή, ε, το Brexit. Πρώτο θέμα λοιπόν, οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Ε, ζητώ συγγνώμη που είναι τόσο ε, μικρά τα γράμματα στις διαφάνειες, αλλά ε, θα σας μιλήσω για αυτές. Εάν κοιτάξετε λοιπόν οποιαδήποτε ανακοίνωση πάνω στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, θα διαβάσετε πόσο αυξάνουν τις εξαγωγές. Εδώ βλέπετε κάποιες δημοσιεύσεις από ανακοινωθέντα τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ε, συμφωνία με την Κορέα, ενώ το δεύτερο απόσπασμα έχει να κάνει με ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στον ε, τομέα της γεωργίας. Και βλέπουμε ότι η συμφωνία με το Μεξικό έχει προσθέσει 105 εκατομμύρια στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νούμερα αυτά όμως δεν μας λένε τι ακριβώς εξάγουμε. Γνωρίζουμε ότι αυξάνεται το εμπόριο. Το εμπόριο σε τι όμως εμπορευόμαστε ευρωπαϊκά προϊόντα, εξάγουμε ευρωπαϊκά προϊόντα ή απλά εισάγουμε προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επανεξάγουμε. Ενώ το ποσοστό των πραγματικά ευρωπαϊκών ε, προϊόντων είναι πολύ χαμηλό. Το ερώτημα που τίθεται εδώ πέρα λοιπόν είναι ποιος ωφελείται από αυτές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και ποια προϊόντα. Όπως ε, μάθαμε από τις ε, παρουσιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ξέρουμε ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου έχουν να κάνουν με προϊόντα που προέρχονται από τους εταίρους. Τι σημαίνει το προέρχονται, σημαίνει ότι έχουν παρασκευαστεί και ότι προσθέτουν αξία στην οικονομία της χώρας αυτής. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, διότι από όλα τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη, Προσπαθούμε να ευνοήσουμε κάποια από αυτά τα προϊόντα περισσότερο, να επιτρέψουμε την εξαγωγή τους σε άλλες χώρες και να επιτρέψουμε η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα από αυτές τις χώρες που να έχουν αρκετή προστιθέμενη αξία από αυτές τις χώρες. Σε ποιο στάδιο λοιπόν αποφασίζουμε ότι αυτό το προϊόν είναι πράγματι ευρωπαϊκό Και πώς αποφασίζουμε ότι αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, ε, ε, συναρμολογήθηκε στην Ευρώπη αλλά δεν προσθέτει αξία στην Ευρώπη άρα ε, δεν ε, θα πρέπει να θεωρείται ευρωπαϊκό. Εδώ βλέπετε μία διαφάνεια, ένα αυτοκίνητο εξάγεται από την Νότια Κορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραίο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο όμως αυτό αποτελείται από πολλά πράγματα. Η μηχανή έχει κατασκευαστεί στη Ιαπωνία, η ε, μηχανή και το σασί είναι από την, ε, οι ρόδες και το σασί είναι από την ε, Κίνα. τα διάφορα τμήματα του αυτοκινήτου προέρχονται από διάφορες χώρες. Πώς λοιπόν καταλήγουμε ότι είναι κορεατικό το αυτοκίνητο και αυτό είναι ένα παράδειγμα αλλά ισχύει για τα πάντα. Το μικρόφωνο ε, στο οποίο μιλώ, ε, το κινητό μου, το κουστούμι μου, η γραβάτα μου. Πώς λοιπόν μπορούμε να αποφασίσουμε ότι αυτό το προϊόν είναι ευρωπαϊκό ή κορεάτικο αντίστοιχα. Αυτά όσον αφορά τις εξαγωγές. Ήδη λοιπόν ανέφερα ότι μπορεί να αποτελείται από διάφορα τμήματα που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορα τμήματα. Το ίδιο ισχύει όμω και για τι εξαγωγέ μα. Να σα δώσω ε, δύο παραδείγματα δύο διαφορετικών μεθόδων ε, ε, κατασκευή οι κανόνες καταγωγής στις ε, συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου μας ε, αποφασίζουν ποιες ευρωπαϊκές χώρες εποφελούνται. Εγώ έχω εργαστεί πολύ στη χημική βιομηχανία, από εκεί λοιπόν θα πάρω και τα παραδείγματά μου. Βλέπετε εδώ τη Βραζιλία και την Κένια, είναι χώρες με τις οποίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Και βλέπετε εδώ την Ρωσία, αγοράζουμε ε, ε, αέριο από την, ε, φυσικό αέριο από την Ρωσία, το οποίο γίνεται αμμόνιο, κατόπιν γίνεται νητρικό αμμόνιο που είναι λίπασμα, το οποίο εξάγουμε. Εισάγαμε φυσικό αέριο ε, και το έχουμε μετατρέψει σε αμμονία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει γίνει νητρικό αμμόνιο, το έχουμε ε, αναμίξει με άλλα πράγματα και έτσι έχουμε καταλήξει σε ένα λίπασμα. Αυτή είναι η μια επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να εισάγουμε το λίπασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην ασχοληθούμε λοιπόν ούτε με το ε, φυσικό αέριο και την αμμονία. Εισάγουμε το λίπασμα, το αναμειγνύουμε με δολομίτη για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξάγουμε αυτό στη Βραζιλία. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές διαδικασίες. Όπως βλέπετε, η πρώτη επιχείρηση έχει ε, εργοστάσιο παραγωγής ε, νητρικού αμμονίου στην Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει. Έχουμε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ε, θέλουμε να τις βοηθήσουμε και τις δύο. Αλλά το θέμα είναι βοηθάμε και τις δύο εξίσου ή βοηθάμε μόνο την πρώτη ή μήπω δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και απλά θέλουμε να τις βοηθήσουμε όλες. Και ε, εδώ τίθεται και το θέμα τη τιμής, διότι καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία που εισάγει λίπασμα από τρίτη χώρα μάλλον έχει πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ε, αν ε, λοιπόν επιδοτήσουμε και τη μία και την άλλη ή αν βοηθήσουμε και τη μία και την άλλη η μία θα ωφεληθεί περισσότερο. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, διότι είπαμε θέλουμε να εισάγουμε αυτοκίνητα που αποτελούνται από τμήματα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι το ένα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις δικές μας επιχειρήσεις. Ποιες θέλουμε να επωφεληθούν περισσότερο στις εξαγωγικές αγορές. Και εδώ βλέπετε μια γενική διαφάνεια. Συνήθως ε, ακούμε ε, τα περί εμπορικών συμφωνιών. Θα αναφερθώ στην TTIP, διότι έχει συζητηθεί τόσο πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα ε, συζητήσει με τους Αμερικανούς σε τους κανόνες καταγωγής, αλλά αυτό που θα γίνει στην πραγματικότητα είναι ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, λάβουν, ε, θα δεχτούν επισκέψεις από πολλούς ε, ανθρώπους από επιχειρήσεις που όμως λαμβάνουν πολλές πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα από άλλες χώρες ε, βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε τις ε, χώρες στα ανατολικά μας, στα νότια μας, ε, πέρα από τις συνδεδεμένες χώρες και την Μέση Ανατολή. Το ίδιο ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή ισχύει ακόμα η ναύτα. Οι Καναδοί και οι Μεξικανοί λοιπόν συμμετέχουν πολύ στο εμπόριο, καθώς και οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής και κατόπιν έχουμε τους μεγάλους παίκτες, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Με όλα αυτά θέλω να σας δείξω ότι στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μπλέκονται και τα συμφέροντα πολλών άλλων χωρών και όταν καθορίζονται οι κανόνες καταγωγής ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές αλλά και ε, ποιοι είναι οι προμηθευτές τους. Να συνοψίσω λοιπόν ε, τρία διαφορετικά μοτίβα. Διαπραγματευόμαστε με τρίτη χώρα, για παράδειγμα στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και θα θέλαμε εδώ ιδανικά όσο μεγαλύτερο μέρος ε, των προϊόντων τους να προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες, διότι δεν θέλουμε να εισάγουμε προϊόντα με αυτό το καθεστώς από χώρες που να, με τις οποίες δεν έχουμε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Κατόπιν έχουμε Ευρωπαίους κατασκευαστές ε, με προϊόντα που βασίζονται σε πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα από αλλού, τις οποίες θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε. Για τις δικές μας επιχειρήσεις λοιπόν, θα θέλαμε ε, σχετικά χαλαρούς κανόνες καταγωγής. Έχουμε όμως και τις ε, δικές μας επιχειρήσεις που πληρώνουν φόρους στην Ευρώπη, επενδύουν στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ βαριά βιομηχανία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επιχειρήσεις που εισάγουν ενδιάμεσα προϊόντα και τους επιτρέπουμε να ξεφύγουν, να παρακάμψουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, για παράδειγμα το σύστημα εμπορίας εκπομπών ή το, την ομοθεσία REACH. Η δεύτερη ομάδα, λοιπόν, βασίζεται σε ε, εισαγόμενα προϊόντα. Και εδώ η λέξη κλειδί και η πολύ κομψή και σύγχρονη διατύπωση ε, είναι η παγκόσμια λυσίδα αξίας ε, και πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλές από τις χώρες αυτές έχουν μεταφέρει τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους σε τρίτες χώρες. Και να σας δώσω ένα ακραίο παράδειγμα πάνω στο οποίο εργάστηκα στο πλαίσιο των ε, διαπραγματεύσεων TTIP. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει ε, μία μέθοδο για την σύμπηξη προϊόντων. Μπορεί λοιπόν ε, κανείς να αναμειγνύει προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα εξάγει ε, χωρίς δασμούς. Βλέπετε εδώ περιπτώσεις όπου λιγότερο από το 15% του κόστους ε, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο κανόνας λοιπόν επιτρέπει σε ένα προϊόν να ονομάζεται ευρωπαϊκό εφόσον μόνο το 15% της αξίας του προσθέθηκε στην Ευρώπη. Ε, το οποίο σημαίνει ότι το 85% της αξίας του προέρχεται από μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας, το δίνω, σας δίνω αυτό το παράδειγμα, διότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι θαμμένες σε ένα παράρτημα ενός πρωτοκόλου μιας ε, συμφωνίας. Ο περισσότερος κόσμος δεν τα βλέπει καν αυτά. Ακούμε τα περί συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, προώθηση των εξαγωγών, αλλά δεν γνωρίζουμε ε, τα στοιχεία που είναι θαμένα στη συμφωνία αυτή. Κανεί δεν βλέπει του κανόνε καταγωγή που του βλέπουν τελικά μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άμεσα ενδιαφερόμενε βιομηχανίε. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που οργανώσατε την σημερινή ακρόαση διότι νομίζω ότι ε, χρειάζεται παρακολούθηση το θέμα αυτό. Για να κλείσω λοιπόν ε, αυτό το τμήμα τη παρουσίαση. γνωρίζετε ότι οι κανόνες καταγωγής είναι πολύ σημαντικοί και καθορίζουν ποιος επωφελείται. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουν να κάνουν ε, με το πρότυπο ανταγωνισμού και ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι διάφορες επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς τρόπους παραγωγής και εάν καθορίζουμε κανόνες καταγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ουσιαστικά λέμε ότι αυτές οι ε, επιχειρήσεις επωφελούνται, ενώ οι άλλες όχι. Αυτό ακριβώς καθορίζουν οι κανόνες καταγωγής. Ποιες ε, παρασκευαστικές διαδικασίες επωφελούνται και ποιες όχι η γενική τάση, και το ανέφερε αυτό ο κύριος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει μια γενική τάση να απελευθερωθούν οι κανόνες καταγωγής. Αν κοιτάξουμε τι γινόταν πριν 10 χρόνια και δούμε τι γίνεται σήμερα, όλο και λιγότερο ευρωπαϊκό περιεχόμενο ε, χρειάζεται για να υποφεληθούν ε, τα προϊόντα από ε, τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Ε, βλέπουμε λοιπόν όλο και λιγότερο ευρωπαϊκό περιεχόμενο στα αγαθά. Και τέλος, πότε-πότε ε, στις ε, διαπραγματεύσεις αυτές σε κάποιοι τομείς της βιομηχανίας υποβάλλουν πολύ ακραίες προτάσεις. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Να αναφερθώ λοιπόν στη διαδικασία. Ποιος αποφασίζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αποφάσει πάνω στου κανόνε καταγωγή, διότι είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα και τόσο δύσκολο που κανένα δεν το καταλαβαίνει. Ακούσαμε εδώ δύο από του πολύ έξυπνους ανθρώπους ε, ε, που γνωρίζουν καλά το θέμα αυτό. Αυτοί οι δύο άνθρωποι και λίγοι ακόμα ε, στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνωρίζουν αυτά. Α, μου τελειώνει ο χρόνο μου, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχα 20 λεπτά στη διάθεσή μου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. 15-20 άνθρωποι εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούνται με το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει πραγματική εποπτεία από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορώ να σα πω ότι είναι γεγονό ότι δεν υπάρχει εποπτεία ούτε από πλευρά των κρατών μελών. Είχα διάφορε συνομιλίε ε, με ειδικού ε, των τελωνίων που συμμετέχουν ε, στην ομάδα του Συμβουλίου για τι εμπορικέ συμφωνίε. Δεν γνωρίζουν τι περιλαμβάνουν οι διαπραγματεύσει και μέχρι να καταλάβει κανεί τι προτάθηκε έχει ήδη συμφωνηθεί με κάποια τμήματα τη βιομηχανία, με τους εμπορικούς εταίρους και το να το αναστρέψει κανείς αυτά είναι αδύνατον. Ε, δύο ακόμα διαφάνειες θα σας δείξω. Εδώ άλλο ένα θέμα που ισχύει γενικά για τις Βρυξέλλες αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και γενικά στους κανόνες καταγωγής είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πού μαθαίνει ποιους κανόνες καταγωγής θα πρέπει να προωθήσει από διάφορες συνομοσπονδίε στις Βρυξέλλε. Και ωραία, εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνομιλεί με τον ε, τομέα του ατσαλιού, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά εντός αυτών των ε, συνομοσπονδιών γίνεται, διεξάγεται ένας πολύ βάρβαρος αγώνας, μια πολύ βάρβαρη διαμάχη και αυτές οι συνομοσπονδίες ε, έχουν πολλά μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι λίγες μεγάλες επιχειρήσεις ε, που δεσπόζουν εντός των νομοσπονδιών αυτών, των συνομοσπονδιών αυτών ε, αποφασίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να προχωρήσω στην τελευταία και πολύ λυπηρή, ε, ε στο τελευταίο και πιο λυπηρό τμήμα αυτής της παρουσίασης, το Brexit, ε, το οποίο απέφυγε να αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι ανησυχούν, αλλά πολλές βιομηχανίες ε, πιστεύουν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελέσει κίνδυνο όσον αφορά την διαμετακόμιση το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παραδοσιακά κράτος ελεύθερου εμπορίου, δεν ε, αγαπάει ιδιαίτερα τον προστατευτισμό και ξέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επικεντρώνεται γενικά στις υπηρεσίες. Ε, θα βλέπουμε λοιπόν επανεξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, τίθεται το θέμα των τελωνίων. Η δυσκολία είναι πώς θα χειριστεί το Ηνωμένο Βασίλειο τις τελωνιακές υπηρεσίες και αν υπάρξει πρόβλημα με τα τελωνία θα υπάρξει και πρόβλημα με την επιβολή των κανόνων. Τελικό στοιχείο λοιπόν, ελπίζουμε να μην καταλήξουμε εκεί. Ακούσαμε όμως τις απειλές για σκληρό Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο να επιδιώξει καθεστώς ε, χαμηλής ρύθμισης, κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα για μας όσον αφορά την επιβολή των ε, κανόνων που ισχύουν για τα τελωνία και τους κανόνες καταγωγής. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο μου. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε, ε, προκλητικά θα έλεγα. Ε, περνάμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Τσερσεύσκα. Um, ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Ευχαριστούμε που καλέσετε και τον ιδιωτικό τομέα σε συζητήσει τέτοιου είδου Πολύ καλή ιδέα. Εγώ προέρχομαι από ακαδημαϊκό περιβάλλον. Συνεργάζομαι και με έναν οργανισμό χαράξης πολιτικής RTH στη Γενέβη, αλλά περισσότερο εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλο ε, εταιριών για όλες τις τελωνιακές ε, πτυχές, ε, ε, αξιολόγηση, κατάταξη της καταγωγής κτλ. Πράγματι, οι κανόνες καταγωγής είναι ένα πολύπλοκο θέμα και αρκετά τεχνικό, οπότε προτιμώ να εστιαστώ σε τρία βασικά θέματα, τα οποία προκύπτουν όταν συζητάει κανείς την καταγωγή. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα 15 λεπτά, δεν το υπόσχομαι, αλλά αν παραλείψω κάτι, υπενθυμίστε μου το μετά. Τα τρία ζητήματα προκύπτουν συχνότερα όταν συζητάμε τους κανόνες καταγωγής στον ιδιωτικό τομέα. Το πρώτο είναι ποιο είναι ο καλύτερος τύπος κανόνων καταγωγής. Το δεύτερο είναι πόσο δύσκολο είναι αυτό για τον ιδιωτικό τομέα. Και το τελευταίο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε το σημερινό ε, σύστημα κανόνων καταγωγής, να το αλλάξουμε, να το τροποποιήσουμε στο μέλλον. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι ποιος είναι ο καλύτερος τύπος κανόνων καταγωγής. Κάτι που ακούγεται πολύ αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του Brexit. Ε, να προσθέσω ότι εργάζομαι στο Λονδίνο, οπότε το Brexit ε, μας απασχολεί στις δραστηριότητές μας. Είναι δύσκολο το ερώτημα. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση από τον ιδιωτικό τομέα. Διαρκώς λέμε ότι κάθε χώρα έχει το δικό της μοντέλο κανόνων καταγωγής. Η ε, υπογράφουν FTA με παρόμοιους τύπους κάνουν καταγωγής, η Ευρώπη όχι. ε, ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσει από αυτή την αρχή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας τύπος είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Και μετά τίθεται το ζήτημα της, προ, του κατά πόσο προστίθεται αξία και χρησιμοποιούνται τέτοια κριτήρια ή πρέπει να χρησιμοποιηθούν κριτήρια ταξινόμησης. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε ορισμένες περιοχές της Ασίας ε, το ζήτημα της προσθήκης αξίας είναι πιο δημοφιλές. Σε άλλες χώρες όπως την Αυστραλία οι περισσότεροι κανόνες καταγωγής ε, έχουν μετατραπεί στην, ε, και εστιαστεί στην κατάταξη. Δεν υπάρχει μια οικουμενική συμφωνία για το ποιο είναι το καλύτερο είδος κανόνων από άψη του ιδιωτικού τομέα. Αν δούμε κάποιες συγκεκριμένες βιομηχανίες και εκεί υπάρχει διαφωνία το συζητήσαμε, είχαμε τις προσπάθειες lobbying από τις διάφορες εταιρείε του ιδιωτικού τομέα και το βασικό θέμα εκεί είναι ότι ακόμη και αν δει κανείς την αυτοκινητοβιομηχανία ή τη βιομηχανία χημικών, η αυτοκινητοβιομηχανία προτιμά την προσθηκη αξίας για την ευκολότερη, ενώ η χημική βιομηχανία προτιμά αλλαγή της καταταξής διότι είναι ευκολότερο αλλά ουσιαστικά εξαρτάται από την αλυσίδα αξίας της κάθε, του κάθε τομέα και μιλήσαμε για το ποιο υποφελείται από αυτού του κανόνε καταγωγή, έχουν σχεδιαστεί να αποτελούν μη δασμολογικό φραγμό, να προστατεύουν την ιστορική αγορά, αλλά αν είναι υπερβολικά αυστηροί, τότε τα επίπεδα χρήση ε, ε, μειώνονται και τα ωφέλη ε, μιας συμφωνίας ελευθερών συναλλαγών ε, δεν επιτυγχάνονται. Περνάω στο δεύτερο ερώτημα, πόσο δύσκολο είναι για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ερώτημα ε, όσον αφορά εσάς οι κανόνε καταγωγής συχνά αναφέρονται από τις εταιρείες ως βασικότατος φραγμός του διεθνούς εμπορίου. Εγώ θα έλεγα ότι πολύ συχνά, παρότι ονομάζονται κανόνες ε, καταγωγής, δεν είναι οι ίδιοι κανόνες καταγωγής που δημιουργούν το πρόβλημα. Είναι το ευρύτερο καθεστώς κανόνων καταγωγής. Σε τι αναφέρομαι, στο διοικητικό γραφειοκρατικό φόρτο και στο σχετικό κόστος συμμόρφωσης με τους κανόνες καταγωγής και για την απόδειξη των κανόνων καταγωγής ε, και οι σχετικές ποινές και οι κίνδυνοι. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αν το κόστος συμμόρφωσης με τους κανόνες καταγωγής είναι υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με το προτιμησιακό ε, ε, Κέρδο που θα επιτύχει μια εταιρεία στο πλαίσιο μιας ε, συμφωνίας ελευθερών συναλλαγών δεν θα το προτιμήσουν, διότι δεν θα έχει πλεονέκτημα. Το βασικό πρόβλημα κατά την απόψή μου είναι ότι το σημερινό καθεστώ κανόνων καταγωγή δεν είναι προσαρμοσμένο στις παγκόσμιες αλυσίδε αξιών. Ε, δεν είναι προσαρμοσμένο στην κατακαιρματισμένα δίκτυα παραγωγής, ε, στα πολύπλοκα μοντέλα παραγωγής, ε, στην κατακαιρματισμένη παραγωγή. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί ε, από πλευρά εισαγωγής και εξαγωγής για την εξαγωγή, το να λάβει κανείς τα έγγραφα καταγωγής, ποιος μπορεί να δράσει ως εξαγωγέας, πώς μπορεί να λάβει το καθεστώς εξαγωγέα και για την εισαγωγή. Υπάρχει, για τις εισαγωγές υπάρχει κάτι άλλο η συνοχή των εγγράφων. Πρέπει να υποβάλει κανείς πολλά έγγραφα για να αποδείξει ε, την καταγωγή, την ε, να... να δώσει εμπορικά έγγραφα, έγγραφα μεταφοράς και όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε εταιρείες διαφορών μεγεθών. Είναι πρόβλημα για τις πολυεθνικές αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα δύο πιο συνήθι παραδείγματα που τα αποδεικνύουν όλα αυτά είναι οι κανόνες ε, απευθεία αποστολή και απευθεία τιμολόγηση. Η απευθείας αποστολή υπάρχει στις περισσότερες ε, ε, FTA. Αποτελεί απέτηση για την εξαγωγή ενό προϊόντος από τη χώρα Α στη χώρα Β άμεσα ώστε να υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση. Σε πολλές περιπτώσεις η μεταφόρτωση είναι δυνατή υπό συνθήκες Φυσικά υπάρχει η προϋπόθεση να μην ακολουθήσει περαιτέρω μεταποίηση και έχουμε και τον έλεγχο των τελωνιακών αρχών. Αλλά το πρόβλημα είναι πώ το αποδεικνύει κανεί αυτό. Πώ αποδεικνύει κανεί τι νοτιοκορεατικές τελωνιακέ αρχέ, ότι ε, τα προϊόντα που μεταφορτώθηκαν μέσω Σιγκαπούρη και πέρασαν κάποιο καιρό στη Σιγκαπούρη διατηρήθηκαν υπό έλεγχο των τελωνίων. Με ποιο έγγραφο μπορεί να το αποδείξει κανεί αυτό και, αυτό και το βασικό πρόβλημα είναι ότι ε, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από τις, διαφο από τις τοπικές αρχές και αυτό είναι πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι δεδομένου του όγκου των εξαγωγών τους πολύ συχνά δυνατούν να γεμίσουν ένα εμπορευματοκιβώτιο. Συχνά τα προϊόντα τους ανασυσκευάζονται ή ε, κάνουν κάποια στάση κάπου ε, καθοδόν. Και το άλλο πρόβλημα είναι η άμεση τιμολόγηση. Πρόβλημα κυρίως για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ε, με περίπλοκο ε, λειτουργικό μοντέλο. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση όπου ένα αγαθό εξάγεται απευθείας από τη χώρα Α στη χώρα Β αλλά βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου υπάρχει μια σειρά χρηματοοικονομικών ε, κίνησεων, δηλαδή τιμολογίων που καλύπτουν αυτή τη μετακίνηση. Υπάρχει ένα βασικό μοντέλο όπου υπάρχουν διάφορες σχετιζόμενες ή όχι εταιρείε και μπορεί να έχει κανείς τρία ή τέσσερα τιμολόγια που να καλύπτουν αυτή την εξαγωγή, αυτή την κίνηση αγαθών. Και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν διατάξεις στο πλαίσιο μιας FTA που να επιτρέπουν αυτή την τιμολόγηση τρίτου μέρους ή αυτή την έμεση τιμολόγηση. Οπότε και εκεί ε, έχει κανείς μια κατάσταση όπου όταν ένα αγαθό ε, φτάνει στον προορισμό του και οι τελωνικές αρχές της χώρας εισαγωγής λαμβάνουν ένα τιμολόγιο από μια χώρα η οποία μπορεί να μην είναι μέρος της ε, Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών. Πώς αποφασίζουν σε αυτή την περίπτωση αν υπόκειται στις ε, απαιτήσει όχι, ε, σε απαιτήσει καταγωγής. Άλλο ζήτημα είναι ότι συχνά ένα τέτοιο εγγραφό περιλαμβάνει εμπιστευτικέ εμπορικέ πληροφορίε που δεν θέλει κανεί να δώσει στου προμηθευτέ του Οπότε μερικέ φορέ ε, δεν είναι καν εφικτό να δώσει τέτοιε πληροφορίε και τέτοια τιμολόγια μια επιχείρηση, διότι περιέχουν ευαισθητέ πληροφορίε. Ενώ λοιπόν οι κανόνε καταγωγή ε, είναι σαφώ καθορισμένοι στο κείμενο μια συμφωνία, οι διατάξει αυτέ ε, συχνά δεν καθορίζονται. Και όπως είπα, το πρόβλημα τελικά πρέπει να απολυθεί από τις τοπικές τελωνιακές αρχές ε, στην χώρα που παρέχει και που ε, είναι δικαιούχος του προτιμησιακού καθεστώτος. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα με το σύστημα ε, κανόνων καταγωγής αυτή τη στιγμή, διότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν ένα τρίτο φραγμό στο εμπόριο. Έχουμε τον πρώτο φραγμό που είναι οι δασμοί που έχουν σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό, μετά έχουμε τον δεύτερο φραγμό οι ίδιοι κανόνε καταγωγής και μετά έχουμε τον τρίτο φραγμό που είναι οι πρακτικές πτυχές ε, της λειτουργίας σε ένα προτιμησιακό καθεστώς. Το πρόβλημα είναι ότι τα, οι πρώτοι δύο φραγμοί ε, ε, έχουν δημιουργηθεί εσκεμένα ε, τέσσερα το αντικείμενο διαπραγμάτευση διάστηκαν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο τρίτος φραγμός δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Είναι απλά ένα πρόβλημα διοικητικό, διότι παρεμποδίζει επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για προτιμησιακή μεταχείριση από το να έχουν πρόσβαση στα ωφέλη μια ε, συμφωνία ελευθερών συναλλαγών. Για όλου αυτού τους λόγους είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι πληροφορίε για το τι ποσοστό του εμπορίου διέρχεται από αυτή τη διαδικασία και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Από τι εμπειρίε του ιδιωτικού τομέα όμω είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό για πολλέ εταιρείε και επηρεάζει τόσο τι μεγάλε όσο και τι μικρέ. Με την αλλαγή λοιπόν των επιχειρησιακών μοντέλων των αλυσίδων ε, προμηθειών ε, πρέπει να προσαρμόσουμε και του κανόνε καταγωγή και το σχετικό μοντέλο. Και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα έχουν κάνει πολλή δουλειά για το θέμα αυτό. Έγιναν διαβουλεύσει με τον ε, ιδιωτικό τομέα, γίνονται όταν διαπραγματεύεστε FTAs για παράδειγμα με το Μεξικό. Αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειε στον τομέα αυτών. Αν οι κανόνε είναι σαφέστεροι, τότε είναι καλύτερη η υλοποίηση και μεγαλύτερα τα οικονομικά ωφέλη. Το θέμα δηλαδή είναι να δίνει κανεί καλύτερη καθοδήγηση στι ελληνικέ αρχέ τη χώρα, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε στο πλαίσιο επιτροπών ε, συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών ή σε πολυμερέ επίπεδο, αλλά απαιτούνται καλύτερη καθοδήγηση των τελωνιακών αρχών. Και μετά τέλο θα σα μιλήσω για του πιθανου τρόπου ε, αναθεώρησης ενδεχομένων των κανόνων καταγωγή ε, στο μέλλον. Δεν θα σας δώσω, θα σας παραθέσω όλα τα στοιχεία, απλά να σας πω πώς θα μπορούσαμε να τους ε, επανεπινοήσουμε τους κανόνες καταγωγής για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από αυτούς και να τους κάνουμε πιο λειτουργικού. Το πρώτο θέμα είναι η ισόρευση, την οποία συζητήσαμε εκτενώς σήμερα το πρωί, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά από την άποψη μιας εταιρεία η ισόρευση επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, κάτι καλό. Αυξημένη ευελιξία ποτέ δεν κάνει κακό. συχνά όταν μιλάμε για συμφωνίες μεγάλων περιφερειών όπως TTIP ή TTP τα ωφέλη μεγάλα. Ξέρουμε ότι αυτές οι μεγάλες συμφωνίες αυτή τη στιγμή ε, δεν γίνουν ιδιαίτερα και να δούμε πόσες θα επιβιώσουμε στα επόμενα χρόνια και τι θα γίνει με αυτές τις ε, εκτενείς συμφωνίες αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι ε, χρήση των σωρεύσεων χωρίς την υπογραφή μεγάλων διεθνών συμφωνιών. Η παραδοσιακή σώρευση χαρακτηρίζεται από δύο βασικούς κανόνες. Ο πρώτος είναι ότι όλες οι χώρες πρέπει να συνδέονται με μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και η άλλη πτυχή είναι ότι αυτές οι FTA πρέπει να περιλαμβάνουν ε, κανόνε καταγωγή ίδιους. Αυτό είναι πρόβλημα, διότι για να έχουν όλες οι FTA οι ίδιους κανόνες ε, τότε ε, παρεμποδίζεται η καινοτομία και οι νέε προσεγγίσει των κανόνων καταγωγή. Ουσιαστικά απαιτείται από τα μέρη να υπογράφουν τους ίδιους τύπους κανόνων καταγωγής και να δεσμεύονται με αυτούς ξανά και ξανά. Αυτό δεν είναι καλό, διότι δεν επιτρέπει να δοκιμάσει κανείς νέες προσεγγίσεις. Μία λύση θα μπορούσε να είναι αυτό που ονομάζουμε ε, εκτεταμένη ισόρευση ή ισόρευση τρίτων μερών. Δεν χρησιμοποιείται πολύ αυτή τη στιγμή. Αναφέραμε κάποια παραδείγματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες για παράδειγμα αλλά υπάρχουν παραδείγματα ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών διμερών όπου αυτό εφαρμόζεται κατά τομέα και ενδεχομένως θα μπορούσε να επεκταθεί στο μέλλον. Ένα παράδειγμα θα ήταν ε, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Καναδά και Κολομβία ή Καναδά και Χιλή, όπου επιτρέπεται η χρήση εξαρτημάτων αυτοκινήτων από τη ΣΥΠΑ και ω καταγόμενων υλικών, δηλαδή το προϊόν πρέπει να εισαχθεί από τη ΣΥΠΑ ή το Μεξικό που δεν ε, είναι μέρος της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών στην επικράτεια τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών και αντιμετωπίζεται σαν να ήταν τα μέλη ε, της, σαν ήταν τα μη μέλη της FTA, μέλη της FTA. Σαν, ε, ενώ δεν έχουν υπογράψει αυτούς τους κανόνες καταγωγής τα μέρη αυτά. Έτσι επεκτείνεται κατά κάποιο τρόπο η περιοχή ισόρευσης χωρίς να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται ενιαία σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένω να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον η εκτεταμένη εκδοχή, ενδεχομένως και στο πλαίσιο του Brexit, ανάλογα με το τι θα γίνει εκεί και κατά πόσο τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποφασίσει ε, να παραμείνει ε, στην Πανευρωπαϊκή ε, Μεσογειακή Ζώνη ή όχι. Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να αναφέρω είναι ο ξυγχρονισμό ή η επικαιροποίηση των κανόνων καταγωγή βάσει νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων. Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για του κανόνε καταγωγή αλλά και για άλλους τελωνιακούς τομείς, για την αξιολόγηση, για την κατάταξη. Εδώ μιλάμε κυρίω για προϊόντα που περιλαμβάνουν υπηρεσίες, νέα προϊόντα πληροφορικής. Στο χώρο της πολιτικής ε, αυτά αναφέρονται ως κινητές ε, ε, εμπορικές υπηρεσίες. Είναι κάτι που συναντάμε πολύ στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, απόψη πελάτη. Πώς αντιμετωπίζει κανείς ένα μηχάνημα παρακολούθησης της ε, φυσικής κατάστασης, ε, πώς το αντιμετωπίζει κανείς αυτό μετρά και τη, ε, την πίεση, αν συνδέεται με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύει, αν συνδέεται με άλλες συσκευές. αυτό το ζήτημα προϊόντων που υπερβαίνουν την παραδοσιακή περιγραφή του προϊόντος υπάρχουν εδώ και καιρό. Πριν δύο χρόνια συζητήσαμε όταν ήρθαν οι, ε, οι μικρές κάμερες, οι μίνι κάμερες που μεταφέρει κανείς μεταξύ του, ε, τι είδους προϊόν ήταν αυτό. Η ποσότητα διασυνδεδεμένων αγαθών με υπηρεσίες θα συνεχίσει να αυξάνεται. Πρέπει να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε αυτά τα αγαθά αλλά και οι κανόνε καταγωγή θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Γιατί αν δούμε την προσθήκη αξία, πώ υπολογίζεται η προσθήκη αξία σε προϊόντα όπου η υπηρεσία αποτελεί τόσο μεγάλο κομμάτι τη αξία. Και αν το προϊόν αυτό καθεαυτό, ε, το μηχανικό κομμάτι είναι πολύ μικρό ε, όσον αφορά την καταγωγή του, αλλά η υπηρεσία που παρέχει είναι πολύ ευρύτερη, είναι καταγόμενο υλικό. Δεν είναι Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα χρειαστεί να, να αντιμετωπίσουμε αργά ή γρήγορα, διότι λαμβάνουμε πολλά ερωτήματα για το θέμα αυτό από τον ιδιωτικό τομέα. Για να συνοψίσω τώρα, οι κανόνες καταγωγής και το τι προετοιμάει ο ιδιωτικός τομέα εξαρτάται από την αλυσίδα ε, προμηθειών. Είναι δύσκολο να πει κανεί τι είναι καλύτερο για κάθε τομέα τη βιομηχανία, αλλά το βασικό ζήτημα είναι ότι οι κανόνε καταγωγή επηρεάζουν διάφορα κομμάτια μια αλυσίδα προμηθειών, διάφορα κομμάτια τη οικονομία μια κοινωνία και πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά πριν την εφαρμογή του γιατί έχουν σημαντικέ επιπτώσεις στο δεύτερο που για μένα είναι το σημαντικότερο κομμάτι αυτή τη παρουσίαση. δεν δημιουργούν πρόβλημα απαραίτητα οι κανόνε καταγωγής αυτή καθεαυτή, αλλά ο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συμμορφωθούν με αυτούς οι εταιρείε από καθαρά πρακτική άποψη. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και το τρίτο θέμα είναι ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο να επεκτείνουμε τον τρόπο χρήσης των κανόνων καταγωγής αυτή τη στιγμή χωρίς να υπάρχει ένα μοντέλο για όλες τις περιπτώσεις και μια απέτηση να είναι πιο ολοκληρωμένη ε, και πιο ευέλικτη για το μέλλον. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ να απαντήσω τις ερωτήσεις. Ε, αν ε, είπα κάτι, αν έφερα κάτι πολύ γρήγορα, μην διστάσετε να με ρωτήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Πιέζει ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, σύντομα. Όχι. Όχι. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε, Πρόεδρε. Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά για τα διάφορα σωματεία. Νομίζω ότι είναι περίπλοκο το θέμα της διαφάνειας έτσι κι αλλιώς, αλλά εμείς δίνουμε διαφάνεια και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και στο Γενικό Κοινό, όπως κάνουμε και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν εμπορικές διαπραγματεύσεις. Όντω υπάρχουν, ε, υπάρχει ολόκληρος κατάλογος κανόνων καταγωγής για τα προϊόντα αλλά και δασμών ε, για τα προϊόντα και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι ενήμεροι. Οι συζητήσεις που γίνονται για την εμπορική πολιτική και τους κανόνες καταγωγής ισχύουν για μεγάλα προϊόντα Τώρα, οι κανόνες καταγωγής δεν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα από ρυθμιστική άποψη. Γιατί μπορεί να έχει προέλευση από την Κορέα, για παράδειγμα, ή όχι. Μπορεί να υποφελείται από προτιμησιακή ε, προτίμηση, όχι, αλλά το REACH εφαρμόζεται έτσι κι αλλιώς. Επ' αυτού πρέπει να είμαστε σαφείς. Οι κανόνες θα ισχύουν όσον αφορά την ασφάλεια και τις προδιαγραφές αυτά εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από την πρόληψη του προϊόντος. Οι κανόνες αυτοί πάντως σίγουρα είναι ένα περίπλοκο ζήτημα τεχνικά μιλώντας. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ωραίο. Είμαι πεπισμένος λοιπόν για τις ε, συζητήσεις αυτές και ότι θα συνεχιστούν ο συγητής μας βέβαια θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θέλω να πω δύο λόγια για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Να ξεκινήσουμε κάτι προφανές. Οι κανόνες καταγωγής καθορίζουν την προέλευση του προϊόντος για εμπορικούς σκοπούς. Και οι περιορισμοί έχουν να κάνουν με την πηγή προέλευσης. Οπότε μόνο τα προϊόντα τα οποία καλύπτουν τους κανόνες καταγωγής έτσι όπως αναφέρονται σε συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες εποφελούνται από την προτιμησιακή μεταχείριση. Από τους κανόνες, για παράδειγμα, των ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, άλλα προϊόντα εποφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση και άλλα όχι και στον ΠΟΕ, στην ομιλία που ακούσαμε τον Ιούνιο του 2017, ακούσαμε για τους προτιμησιακούς κανόνες σαν έναν τομέα ζωτικής σημασίας. Και γιατί, γιατί καθορίζουν τις συμφωνίες τις εμπορικές και τις καταστούν πιο περίπλοκες και πιο πολυεπίπεδες. έχουμε πάρα πολλές εμπορικές συμφωνίες ανά τον κόσμο. Και τώρα το ζήτημα είναι, εποφελούμαστε από αυτούς τους κανόνες καταγωγής ή ποιος τελικά εποφελείται. Αποτελούν εσωτερικό τμήμα των διαπραγματεύσεων και προνόμιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. κοιτάξτε την αίθουσα. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Θα έπρεπε να αλλάξει αυτό. Πάντως στα πλαίσια των γενικών συζητήσεων για τα ωφέλη από το ελεύθερο εμπόριο, οι κανόνες καταγωγής είναι πάρα πολύ επίκαιροι. Γιατί έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το οποίο δεν είναι λίγη ευτυχία στον κόσμο. Ποιος τελικά υποφελείται από το ελεύθερο εμπόριο. Ακούσαμε πολλά για την ανάγκη αναρμόνισης των κανόνων καταγωγής και ότι θα έπρεπε στην πράξη να είναι πιο εύχρηστη. Καλός ο στόχος. Συγχρόνως όμως πρέπει να προσέξουμε να μην αποδυναμωθούν υπερβολικά. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι υπάρχει και το θέμα των εσόδων, γιατί έχουμε τους τελωνιακούς δασμούς που αποτελούν μέσω εσόδων αν μειωθούν, διευκολύνεται μεν το εμπόριο, αλλά μειώνονται τα έσοδα. Οπότε πρέπει να εφαρμόσονται σωστά οι κανόνες καταγωγής, γιατί επηρεάζουν, όπως είπαμε, όχι μόνο το εμπόριο, αλλά και τα έσοδα μιας χώρας. Επίσης, για τους κανόνες καταγωγής, χρειαζόμαστε να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο. Όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν ε, μια ιδιαίτερα περίπλοκη αλυσίδα αξίας. Μπορεί να είναι καλό ή κακό αυτό, πάντως στη σημερινή οικονομία και τους κανόνες καταγωγής γίνονται πολλές διευθετήσεις. Να έχουμε υπόψη μας ότι για να καταλάβει κανείς αυτόν τον ε, τομέα και να τον ε, αντιμετωπίσει, πρέπει να φροντίσει να μην έχει αρνητικές συνέπειες από αυτού. Να μην τον αλλάξει δηλαδή προς το χειρότερο. Και το Brexit ε, φυσικά μας απασχολεί. Να είμαστε πιο προσεκτικοί ανάλογα με την κατεύθυνση που θα πάρουν τα πράγματα τελικά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαιτήσουμε αυστηρούς κανόνες καταγωγής στην Συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου Ευρώπης, ώστε τα αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι όντως αγαθά Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι, αυτό. Είναι πολύ απλό. Αλλιώ συμφωνώ με αυτά που είπαν οι ομιλητέ ότι το θέμα των προτιμησιακών κανόνων καταγωγή ήταν κάτι που είχε μείνει κάτω από το χαλί για πολύ καιρό. Και ότι πρέπει να ρίξουμε λίγο φω σε αυτού και να συμμετέχει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για τους κανόνες καταγωγής θα έχουμε περισσότερους ευρωβουλευτές παρόντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε το σύστημα. Μερικές φορές έχουμε κατώτατο όριο δασμών 3% και μπορούμε να σκεφτούμε εάν θα πρέπει σε όλα τα προϊόντα να εφαρμόσουμε ε, αυτό το καθεστώς. Ε, αλλιώς ε, θα είναι υπερβολικό το γραφειοκρατικό άχθος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την πρόκληση της ψηφιοποίησης καθώς και τις νέες διαχωριστικές γραμμές, πότε μιλάμε για προϊόν, πότε μιλάμε για υπηρεσία κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ και ε, τους ακροατές μας. Θα τα πούμε σύντομα, επόμενη συνάντηση ε, θα πραγματοποιηθεί στις 11 και, 10, και κατόπιν στις 30 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.